συγκεκριμένα την κατάσταση στο Ιράκ. Παρακαλώ κύριε Ντελαβέντοβα. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αξιότιμοι κύριοι Ευρωβουλευτές. Η κατάσταση στο Ιράκ, όπω γνωρίζετε, είναι πάρα πολύ σοβαρή και τα απορίσματα του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων του Ιουνίου εκφράζουν τη βαθιά ανησυχία τη Ευρωπαϊκή Ένωση, καταδικάζοντα τι επιθέσει στι οποίε προέβη το Ισλαμικό κράτο του Ιράκ και τη Ανατολή, το Ισλ. Ε, στο Ιράκ έχει ξεσπάσει μια ε, επανάσταση των Σουνιτών, όχι μόνο από το ΙΣΙΛ, αλλά και από διάφορες άλλες ένοπλες δυνάμεις, μεταξύ των οποίων νέο ε, μπαθ και φιλετικές ομάδες. Το ΙΣΙΛ μαζί με διάφορους ένοπλους μαχόμενους αντιπροσωπεύει μια πιο άμεση απειλή στο Ιράκ από ό,τι στη Συρία. Μια τέτοια οργάνωση με ξένους μαχητές που κατατάσσονται αποτελεί ένα πραγματικό κίνδυνο για του γείτονε του Ιράκ, όπω ο Λίβανο και η Ιορδανία, αλλά και για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η επιδείνωση τη κατάσταση ασφάλεια στο Ιράκ απορρέει από παράγοντε τόσο εσωτερικού όσο και εξωτερικού. Χωρί αμφιβολία, η κρίση στη Συρία επέτρεψε στο Ίσιλ να μπορέσει να αποκτήσει στην περιοχή μια βάση και ένα σημείο κίνηση για τη δημιουργία του αποκαλούμενου Ισλαμικού κράτου σε Συριακά και Ιρακινά εδάφη. Ωστόσο τα αίτια της πρόσφατης ε, αναταραχής δεν περιορίζονται στην έκφραση μιας δρομοκρατικής ιδεολογίας. Ε, τα αίτια των μεγαλύτερο μέρος των ένοπλων μαχητών βασίζονται στην δυσαρέσκεια που δρέφει η κοινότητα των Σουνιτών εδώ και πάνω από 10 χρόνια απέναντι στην Ιρακινή κυβέρνηση την οποία κυριαρχούν οι ΣΥΤΕΣ. Ανάμεσα στα αίτια για τη δυσαρέσκεια είναι η αυθαίρετη εφαρμογή από πλευρά της κυβέρνησης του Ιράκ πολιτικών αποβαθοποίησης, δηλαδή απομάκρυσης των ε, ε, μελών του ΜΠΑΘ, η ε, αδράνεια να, και η, η αδυναμία να, να καλυφθούν οι βασικές ανάγκες της κοινότητας των Σουνιτών και η παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που γίνεται από τις δυνάμεις της ασφάλειας. Οι διαμαρτυρίες της τοπική, του τοπικού πληθυσμού κατέληξαν σε βίαιες συγκρούσεις ανάμεσα στις αρχές της Ασφάλεια της Ιρακινές, τις οποίες κυριαρχούν οι σύντε και των τοπικών φυλών και τις τοπικές φυλές. Αυτή η κατάσταση έδωσε στο Ισραήλ την ευκαιρία να εγκαθιδρυθεί σε αυτά τα εδάφη, όπως έδειξε η επίθεση που έγινε σε Ιρακινά εδάφη τον Ιούνιο. Η ταχύτητα και αποτελεσματικότητα αυτή τη επίθεση ε, ε, εξέπληξαν τη διεθνή κοινότητα. Όλοι οι πολιτικοί και θρησκευτικοί ηγέτες του Ιράκ συμμερίζονται την ευθύνη για να αντιμετωπίσουν τα αίτια που βρίσκονται στη βάση αυτών των εντάσεων. Η Ιρακινή κυβέρνηση πιο συγκεκριμένα καλείται να παίξει έναν ρόλο μετριοπαθή, αποφεύγοντας τις υπερβολές τόσο στο λόγο όσο και στις πράξεις. Η τραγική απόρρεια αυτών των συνθήκων ε, ε, ε, της ασφάλειας δίνεται από τις ανθρωπιστικές επιπλοκές γιατί σήμερα Συνολικά, δύο εκατομμύρια Ιρακινοί έχουν αναγκαστεί να φύγουν από τα σπίτια του. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει μεγάλε ανησυχίε όσον αφορά την εξέλιξη αυτή τη ανθρωπιστική κρίση και τη μαζική εσωτερική μετακίνηση εξόδου μάλλον των πολιτών που προσπαθούν να φύγουν τι ένοπλες συγκρούσεις. Η Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω της ΕΚΟ μέχρι στιγμής έχει δώσει 12 εκατομμύρια ευρώ για ανθρωπιστική βοήθεια. Πρόκειται για χρήματα τα οποία απευθύνονται στους Σύριους πρόσφυγες και τους πολίτες που έχουν εσωτερικά ε, μετακινηθεί στο Ιράκ. Επιπλέον η Ευρωπαϊκή Ένωση συντονίζει τις δράσεις της με άλλους ε, δωρητές και διεθνείς ε, οργανισμούς και θα ήθελα να επενέσω τις προσπάθειες που καταβάλει η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι διεθνείς οργανισμοί σε, τόσο, σε πολύ δύσκολες τοπικές συνθήκες που οφείλονται στον διασκορπισμό των εσωτερικών προσφύγων σε όλο το έδαφος του Ιράκ. Η Ευρωπαϊκή Ένωση διαρκώς ενημερώνεται για την κατάσταση προσαρμόζοντας τις δράσεις βοήθειας ανάλογα με τις εξελίξεις επιτόπου. Μια άλλη συνέπεια της τρομερής κρίσης που έχει πλήξει το Ιρακινά εδάφη αφορά την περιοχή του Κουρδιστάν. Τις προηγούμενες εβδομάδες το Κουρδιστάν ε, του Ιράκ ανακοίνωσε μονομερός ότι σκοπεύει το φθινόπωρο να προβεί σε δημοψήφισμα όσον αφορά την ανεξαρτησία του. Επιτρέψατε μου να υπογραμμίσω ότι το, Κουρδιστάν, το Ιρακινό Κουρδιστάν είναι ένα πρότυπο σταθερότητα σε όλη την περιοχή και έχει αποτελέσει έναν βασικό συνομιλητή για του διεθνεί ε, συνομιλητέ. ιδιαίτερα ανταποκρινόμενο στην ανθρωπιστική κατάσταση στο Ιράκ. Αυτή η συνεργασία αξίζει να ανταμειφθεί. Ωστόσο θεωρούμε πως οι μονομερείς κινήσεις προς την ανεξαρτησία δεν βοηθούν να ξεπεραστεί η κατάσταση κρίσης στο Ιράκ και θα μπορούσαν να αποτελέσουν ένα κίνδυνο, ένα πρόβλημα για το ίδιο το Κουρδιστάν. Καλέσαμε όλα τα μέρη, τα ενδιαφερόμενα μέρη να διερευνήσουν τη λύση για αυτήν και για άλλες ε, ε, πτυχές στη σύσταση και στο Σύνταγμα του Ιράκ που αν εφαρμοστεί πλήρως μπορεί να δώσει απαντήσεις σε πολλές από τις κουρδικές διεκδικήσεις. Η μετάβαση που ξεκίνησε στο Ιράκ πριν από 10 χρόνια και πάνω και που ανέκαθεν είχε τη στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι δύσκολη διαδικασία. Παρά τις ε, πολλές ε, ε, ε παύσεις στη διάρκεια των ετών και ακόμα και αν και σήμερα οι προπτικές του Ιράκ που επιτέλους έχει μπει σε μια διαδικασία ειρήνευσης και σταθερότητας και απειλείται αυτή η κατάσταση πρόσφατα παρατηρήθηκαν και θετικά στοιχεία. Οι εκλογές της 30 Απριλίου είδαν ε, θρόα προσέλευση στις κάλπες 60% των ε, των ψηφοφόρων παρουσιάστηκαν παρά τις δύσκολες συνθήκε ασφαλείας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έστειλε μια αποστολή ειδικών για να παρακολουθήσουν την εκλογική διαδικασία και να μας αναφέρουν τα όσα έγιναν εκεί. Σύμφωνα λοιπόν με τα πορίσματα των εμπειρογνωμόνων, παρά κάποια προβλήματα και ιδιαίτερα την αποκλεισμό σημαντικού αριθμού ψηφοφόρων Σουνιτών στην επαρχία του Άνμπαρ λόγω της βίας, ε, η εξέλιξη των εκλογών θεωρήθηκε ικανοποιητική. Το ποσοστό συμμετοχή δε στι εκλογέ αυτέ που έγιναν λίγε εβδομάδε πριν από την ε, επανάσταση των Σουνιτών δείχνει τη δέσμευση των Ιρακινών πολιτών υπέρ της δημοκρατίας και της ενότητας στο Ιράκ. Πέρα από την ασφάλεια, σήμερα η πιο άμεση απειλή στο Ιράκ αφορά την ικανότητα των ε, μετριοπαθών ε, πολιτικών ηγετών να προωθήσουν την πολιτική διαδικασία. Αυτό είναι το μήνυμα που στείλαμε σε αυτού του ηγέτε τι τελευταίε εβδομάδε. Ο σχηματισμό ε, μια νέα κυβέρνηση μετά από τι εκλογέ τη 30 Απριλίου είναι θέμα προτεραιότητα. Ο ορισμός του Προέδρου του νέου, συμβου, του, του νέου νέα συνέλευση εχθές 15 Ιουλίου ήταν ένα βήμα στη σωστή κατεύθυνση. Ε, τώρα θα πρέπει να οριστεί ο πρόεδρος της, ε, της Δημοκρατίας για να μπορέσει να οριστεί και ο Πρωθυπουργός και να σχηματίσει η κυβέρνηση. Η νέα κυβέρνηση θα πρέπει να αναζητήσει το διάλογο με όλες τις κοινότητες που συναποτελούν το Ιράκ, συμπεριλαμβανομένες της κοινότητας των Σουνίτων που αυτή τη στιγμή αποκλείεται από την ε, πολιτική διαδικασία. Χωρίς ε, μια καθολική διαδικασία όπου θα συμμετέχουν όλοι και πραγματικό διάλογο η Ιρακινή κοινωνία δεν θα προχωρήσει στη συμφιλίωση. Όπως έχει επαναλάβει η εκπρόσωπος κάθε άστον επανελειμμένα, η ε, έξοδος από την κρίση περνά καταρχήν από μια πολιτική λύση, η οποία θα πρέπει να θέσει τις βάσεις για μια απάντηση και στο επίπεδο της ασφάλειας. Αντίθετα, είναι πολύ πιθανό ε, εξαιρετικά αυστηρά μέτρα ασφαλείας να τροποδοτήσουν τη διχόνοια, την, ε, τη διχόνοια και να, να προκαλέσουν νέα προβλήματα στον πληθυσμό του Ιράκ. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι έτοιμη να παρέμβει με κάθε τρόπο που θεωρείται χρήσιμο για να διευκολυνθεί ο διεθνό διάλογο μαζί με του διεθνού μα εταίρου. Παρά τη σοβαρότητα τη κατάσταση επιτόπου, η Ευρωπαϊκή Ένωση συνεχίζει να δίνει βοήθεια και στήριξη στο Ιράκ όποτε αυτό είναι δυνατό, ιδιαίτερα στο πλαίσιο του σχεδιασμού, τη ενημέρωση μάλλον και της ε, ε, ουσιαστικής βοήθειας στην ανάπτυξη. Αυτό είναι ένα μήνυμα τη μόνιμη ε, προσήλωση και δέσμευση τη Ευρωπαϊκής Ένωσης προς το, υπέρ του Ιράκ, ώστε να προωθηθούν οι δυνατότητες διακυβέρνηση και να στηριχθεί η δημιουργία βασικών υπηρεσιών. Αυτή η βοήθεια συμπεριλάβει και μια ακόμα στήριξη με τα, τα μέτρα προώθηση του κράτου δικαίου για να δοθεί συνέχεια στι εργασίε της αποστολή You Just Lex. Υπό το φως της νέας κατάστασης της ασφάλειας στο Ιράκ, οι ειδικοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης αξιολογούν επίσης πιθανές δυνατότητες στήριξης για τις δράσεις κατά της τρομοκρατίας. Ωστόσο, ο αγώνα κατά τη τρομοκρατίας στο Ιράκ οφείλει να σεβαστεί τι αρχέ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του διεθνού ανθρωπιστικού δικαίου. Η Ευρωπαϊκή Ένωση απορρίπτει την άποψη σύμφωνα με την οποία οι παραβιάσει των ανθρωπίνων δικαιωμάτων είναι το απαραίτητο ή αναπόφευκτο τίμημα της ασφάλειας. Η αναποφευκτο τιμημα τη ασφαλεια η προσπαθεί προσπαθει επιση να προωθεί τη συνεργασία ανάμεσα στα κράτη-μέλη όσον αφορά του ξένου μαχητέ ε, το, με, με, κατόπιν δικού του αιτήματο. Τέλο, η Ευρωπαϊκή Ένωση διατηρεί την προσήλωσή τη υπέρ τη Συμφωνία Εταιρική σχέση και συνεργασία με το Ιράκ και θα συνεχίσει να ε, προωθεί αυτή τη συνεργασία. Σχετικά θα ήθελα να εκμεταλλευτώ την ευκαιρία για να καλέσω τα κράτη-μέλη που δεν το έχουν ακόμα πράξει να ολοκληρώσουν όσο γίνεται πιο σύντομα τη διαδικασία επικύρωση τη συμφωνία. Σα ευχαριστώ για την προσοχή σα. Σα ευχαριστούμε κύριε Ντελαβέντοβα και ξεκινάμε τη συζήτηση. Πρώτο ομιλητή είναι ο Αρνό Ντανζόν. Για δύο λεπτά. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Αργά ξυπνήσαμε και είναι οδυνηρό αυτό Χρειαζόταν αυτή η επέλαση των τζιχαντιστών και η δημιουργία του Ισλαμικού κράτους ε, με την κατάληψη της Μοσούλης για να συνειδητοποιήσουμε αυτή την τεράστια στρατιωτική και πολιτική καταστροφή στο Ιράκ. Μπορούμε ως Γάλλοι, εγώ ως Γάλλος ε, το ε, θεωρώ σχετικά εύκολο, να θυμόμαστε συνέχεια το 2003 το τραγικό λάθος της Αμερικανικής εισβολής στο Ιράκ. Ιστορικά αποδείχθηκε ότι δεν βοήθησε τίποτα, αλλά δεν χρειάζεται ίσως να το αναφέρουμε σήμερα γιατί έκτοτε έχουν γίνει πολλά. Από το 2011 και μετά, σωστά λίγο πολύ νομίζω, έχουμε εστιάσει την προσοχή μα στη Συρία. Αυτό όμω έκρυψε τη σοβαρότητα τη κατάσταση στο Ιράκ. Είναι απλουστευτικό σήμερα, όπω πολύ συχνά ε, ακούμε και διαβάζουμε και το έχουμε ακούσει και εδώ σε αυτή την αίθουσα την επιδείνωση της κατάστασης στο Ιράκ να τη θεωρούμε απλή και μόνο συνέπεια του εμφύλου πολέμου στη Συρία. Η Φαλούτζα ξέρετε, κατελήφθη πριν από έξι μήνες από τους τζιχαντιστές. Οι τζιχαντιστές αυτοί, αυτό ο, Ισλαμική, ο Ισλαμικός στρατός, έχει βαθιές ρίζες στο Ιράκ. Είναι οι περισσότεροι ηγέτες της ε, Ιρακινοί και ευημερούν ε, λόγω της αδιαλαξίας και του σεχταρισμού της Ιρακινής κυβέρνησης που έριξε ε, στις ανοιχτές αγκάλες ε, αυτών των τζιχαντιστών τους Σουνίτες οι οποίοι βγήκαν έφυγαν από την ε, εξουσία και επειδή ο Ιρακινός στρατός που ποτίθεται ότι είναι εκπαιδευμένος και εξοπλισμένος δεν είναι αποτελεσματικός, ε, βλέπουμε ότι ε, έχει πρόβλημα ενώ τα αποθέματα και τα πυρομαχικά και τα όπλα τα καταλυστεύουν οι τσιχαντιστές. Πρέπει να στηρίξουμε μια διακυβέρνηση στην οποία θα συμμετέχουν όλες οι συνιστώσεις της Ιρακινής κοινωνίας. Θα πρέπει να βρούμε μια λύση που θα προασπίζεται την, η, η ακαιρεότητα και πολιτική του Ιράκου και τον κατακαιρματισμό. Ε, είναι ασαφείς οι σχέσεις και το λέω διπλωματικά ε, οι σχέσεις ε, κάποιων Σουνιτών και κάποιων κρατικών και μη κρατικών ε, στρωμάτων στον κόλπο, βλέπουμε απειλές από την κατάσταση αυτή και για τη δική μας ασφάλεια, όχι μόνο για την περιοχή. Επίσης, στις 24 Μαΐου έγινε από τσιχαντιστή Γάλλο αιματοχυσία στο Εβραϊκό Μουσείο των Βρυξελών με δολοφονία τουριστών. Πρέπει και αυτές τις δολοφονίες να μην τις ξεχνάμε. Άννα Γκόμες, τρία λεπτά. Μόλις αρχίζει να ανακτά το Ιράκ ε, τις δυνάμεις του μετά από την Αμερικανική εισβολή του 2003 και επανέρχεται ε, η βία και η βαρβαρότητα μέσω των ε, τρομοκρατικών δυνάμεων του ΙΣΙΣ που διακήρυξαν την ύπαρξη του Ισλαμικού κράτους του Ιράκ και της Ανατολής και συνεχίζουν καταστρέφοντας κληρονομιά και οποιοδήποτε σημείο μοντερνισμού στο Ιράκ. Ε, η κυβέρνηση Αλμαλίκη συνεισέφερε σε αυτή την αποσύνθεση της εθνικής ενότητας, για, ενότητας να δώσει απαντήσεις στα θεμητά αιτήματα των ε, Σουνιτών. Η, ε, η, καταστολή των διαμαρτυριών των πληθυσμών των Σουνιτών από πλευράς των ενόπλων δυνάμεων στο, όπου, όπου βασικά χειρουργούν οι Σίτε στο Άνμπαρ δείχνουν την κατάσταση. Ο Αλμαλίκ έχει μεγάλε ευθύνε. Πρέπει να αποσυρθεί και να δώσει χώρο για το σχηματισμό μια νέα κυβέρνηση. Να δώσει τη δυνατότητα για μεγαλύτερη ασφάλεια. Ξεκινώντα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τη ΕΠΑ, το Ιράν, θα πρέπει να επικεντρώσουμε τι δυνάμει μα ώστε να υπάρξει ένα σταθερό και ενωμένο Ιράκ. Οι εκλογέ τη 23 Απριλίου ε, θα έπρεπε να οδηγήσουν σε αυτή την πορεία. Αυτή θα πρέπει να είναι η προτεραιότητα ε, της Εθνοσυνέλευσης και η δημιουργία και η παροχή μάλλον βασικών υπηρεσιών. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να συνεχίζει να μην αναμειγνύεται πολιτικά στην περιοχή. Θα πρέπει να προωθήσει το διάλογο ανάμεσα σε όλες τις κοινότητες ε, του Ιράκ, ε, ώστε να αυξηθεί η δυνατότητα διακυβέρνησης θα πρέπει να υπάρξει κεντρική προσπάθεια για να σταθεροποιηθεί η κατάσταση στο Ιράκ και να σταματήσει ο πόλεμος στην Συρία. Να ε, σταματήσει αυτό η σύγκρουση ανάμεσα στους Σουνίτες και στους Σιήτες. Ε, και συμφωνώ με τον κύριο Ντανζάν και πράγμα που αναφέρεται και στο αυριανό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, να μιλήσει με τις χώρες του Περσικού κόλπου για να σταματήσουν να στηρίζουν ε, διάφορες ε, ομάδες όπως η Ίσεις και άλλοι που είναι σεχταριστικές και τρομοκρατικές ομάδες. Πρέπει να χρησιμοποιήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση τη Συμφωνία εταιρική Σχέσης και Συνεργασίας για να υπάρξει η συνεργασία εκεί την καταπολέμηση της τρομοκρατίας. να μην απορείτε που όλοι οι Ιρακινοί προσπαθούν να βρουν καταφύγιο και παράδειγμα στο άλλο Ιράκ που λειτουργεί θαυμάσια στην περιοχή του Κουρδιστάν. Η, πρόσφατα, η πρόσφατη πρωτοβουλία για να διοργανωθεί ένα δημοψήφισμα όσον αφορά την ανεξαρτησία του Κουρδιστάν τις τελευταίες εβδομάδες είναι κατανοητή. Ε, όμως ακόμα και μια μονομερής ε, ανεξαρτησία η οποία θα είναι ειρηνική δεν θα λύσει τα προβλήματα. Είναι δυνατόν να αναζητηθούν λύσεις εναλλακτικέ συνταγματικού τύπου για ένα Κουρδιστάν το οποίο θα συνεχίσει να είναι κομμάτι του Ιράκ. Τέλος κύριε Πρόεδρε, ο πόλεμος στη Συρία, κίνδυνος ε, τρομοκρατία στο Ιράκ αλλά και αλλού θα πρέπει να μας κάνουν να καταλάβουμε πως και η ευρωπαϊκή ασφάλεια κινδυνεύει γιατί βλέπουμε χιλιάδες διχαντιστές ευρωπαϊκής προέλευσης να πολεμούν επί τόπου και να επιστρέφουν ε, εκπαιδευμένοι για να ενεργήσουν και στην Ευρώπη. Είναι πολύ σημαντικό γιατί είδατε τι συνέβη στο Μουσείο το Ευρωπαϊκό Μουσείο των Βρυξελών. Έχετε μια μπλε κάρτα, κύριε Γκόμας, τη δέχεστε. Κόντι. Κύριε Πρόεδρε, κυρίε και κύριοι, απλά θέλω να επιστήσω την προσοχή του Κοινοβουλίου σε ένα παράδοξο το οποίο ανέφερε η κυρία Γκόμης και ο κύριος Ντάνζα που από τη μία φράζουν τη θλίψη τους ε, για τις επιπτώσεις ε, της επέμβασης στο Ιράκ ε, που δημιούργησαν αυτές τις συγκρούσεις μεταξύ των και Σουνιτών ξεχνάνε να θυμίσουν όμως ότι στήριξαν τη στρατιωτική επίθεση στη Λιβύη που απο... ακριβώς τα ίδια αποτελέσματα έχει με την διάσπαση της χώρας σε διάφορες φυλές έτοιμα πρέπει, μια ερώτηση πρέπει να κάνετε, όχι παρέμβαση, διακόπτει ο πρόεδρος, τον κύριο Σοπχάντα. Παρακαλώ να απαντήσετε. Με μικρόφωνο κι εσείς παρακαλώ να απαντήσετε. Δεν έχετε δίκιο και δεν πρέπει να συγκρίνουμε τις δύο ε, περιπτώσεις, αν και έχουν βέβαια κάποια κοινά στοιχεία. Εγώ ήμουν στη διάρκεια του πολέμου στη Βενγάζη, στη Λιβύη και είδα τι έκανε η διεθνής κοινότητα. Ουσιαστικά μόνο στήριζε τον ε, λαό που πάλευε κατά ενός δικτάτορα, καταπιεστή. Και κάποιοι είχαν business ε, με αυτόν τον ηγέτη. Μη συγκρίνουμε ανώμια πράγματα λοιπόν. Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Τζαλς Τάνοκ για δυόμιση λεπτά. Κύριε Πρόεδρε, ε, κύριε Μαλακή μα ε, ήταν πρόεδρο τη κυβέρνηση από τότε που έγινε πρωθυπουργό το 2006 και έχει ε, εκμεταλλευτεί τι ε, εντάσει μεταξύ των ε, ΣΥΙΤΟΝ και των ΣΥΝΙΤΟΝ. Το καθεστώς του, του Αλμαλίκη, το οποίο έχει πλειοψηφία από τι τελευταίε εκλογέ 30 Απριλίου, ουσιαστικά και δυστυχώ υποστηρίζεται από το Ιράν και από τι ηγεμονικέ τη τάσει στην περιοχή. Και οι σουνικέ φυλές, αραβικέ φυλέ, υπόκειται διακριτική μεταχείριση και εκατοντάδε χιλιάδε άμαχοι έχουν χάσει τη ζωή του, ιδιαίτερα στην Αλάμπα, στο όνομα της, του πολέμου κατά των τζιχαντιστών της ISIS, Και η σουνητική αραβική κοινότητα και οι υποστηρικτές του Σονταμ Χουσέν αντιμετωπίζουν ε, συμμαχίες ε, με την ίσης για να καταπολεμήσουν τους Κουρδιστά, τις ε, κυβερνητικές δυνάμεις. Και στο Κουρδιστάν πλέον έχουν διαμορφωθεί λοιπόν τρεις ξεχωριστές οντότητες που απειλούν την, την εδαφική ακεραιότητα του Ιράκ. Και έτσι υπάρχει λοιπόν ο κίνδυνος να υπάρξουν συγκρούσεις και στη Συρία σε ό,τι αφορά και τον περσικό κόλπο και την ε, στρατιωτική του εξοπλισμό. Θα πρέπει να σταματήσει όμως η δράση του Αλμαλίκη. Θα πλέον έχει ανακηρυχθεί ως χαλφάτο Ισλαμικό, όπου επικρατεί ε, η βαρβαρότητα του νόμου της Σαρίας και όπου θανατώνονται οι μειονότητες των χριστιανών και στο Ηνωμένο Βασίλειο και στην υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχει ριζοσπαστικοποίηση και αποτελεί αυτό σημαντική, σημαντικό κίνδυνο όταν επιστρέφουν στις χώρες τους. Πρέπει λοιπόν κατεπηγόντως να βρούμε μια λύση και θα πρέπει να κοιτάξουμε και τις περιφερειακές και τις ε, διεθνείς δυνάμεις που μπορούν να μας ε, υποστηρίξουν. Ο κουρτικός ε, στρατός είναι πολύ επιτυχή σε ό,τι αφορά την πράσπιση του Κυρκούκ και σε ό,τι αφορά την πράσπιση των συνόρων και την προστασία των χριστιανικών μειονοτήτων. Το Κουρδιστάν λοιπόν έχει εξαγγείλει τη διεξαγωγή δημοψηφίσματο για τη μονομερή εξαγγελία τη ανεξαρτησία. Είναι πάρα πολύ σημαντικό και αυτό το είχε, υποσχεθεί από τι δυτικέ δυνάμει στη συνθήκη του Σεμπρό το 1920 και τώρα λοιπόν πλέον αυτό ενδεχομένω να καταστεί η πραγματικότητα που δεν μπορούμε να αρνηθούμε. Ευχαριστώ. Μπλε κάρτα. Την αποτέχεστε. Όχι, πρέπει να μας πείτε αν τη δέχεστε. Δεν εξαρτάται από κάποιον άλλον. Εσείς δέχεστε το ερώτημα. Ναι, άμα θέλω να ξέρω από ποιον είναι. Ο κύριος Τζόναθαν Άρνοντ, παρακαλώ. 30 δευτερόλεπτα. No, questo è il regolamento, mi scusi. Ναι, αυτός είναι ο κανονισμός, με συγχωρείτε. Όταν η κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου ανέλαβε δράση για να απομακρύνει τον Σαντάμ Χουσέιν, ήταν περίεργα και αντιφατικά τα μηνύματα. Καταρχά, ε, όπλα μαζική καταστροφή, τρομοκρατία και προστασία των ερακινών. Ε, συμφωνώ ότι ήταν κακή, κακό ο σχεδιασμό τη κυβέρνηση ε, Μπλερ και ότι η στρατιωτική παρέμβαση ποτέ δεν θα έπρεπε να έχει λάβει χώρα και ποτέ δεν θα πρέπει να λαμβάνει η χώρα εάν δεν υπάρχει κάποιο σαφή στρατιωτικό στόχο. Συμφωνείτε. Απάντηση. Συμφωνώ ότι η κυβέρνηση Μπλερ τότε ήταν μάλλον ε, λακωνική σε ό,τι αφορά την αλήθεια και ότι και εμείς ε, και εγώ που είχα υποστηρίξει τότε τον πόλεμο, αν ήξερα τότε αυτά που ξέρω τώρα, ενδεχομένω να είχα τελειώσει διαφορετική στάση. Αλλά συμφωνώ ότι η παρέμβαση στο Ιράκ, η οποία είχε καλέ προθέσει και ότι ήταν ανθρωπιστική, έχει, ε, έχει τελικά καταλήξει μια δεκαετία αργότερα σε μεγάλο χάο και καταστροφέ Άλλη μια αίτηση για μπλε κάρτα δεν έχετε κύριε Τάνοκ. Κοιτάξτε, είναι η πρώτη φορά σε 15 χρόνια που ο άνθρωπος που βρίσκεται στην Προεδρία είναι, δεν μας λέει από ποιον προέρχεται αυτή η ερώτηση. Πρέπει κανείς να γνωρίζει ποιος ε, έχει σηκώσει η μπλε κάρτα. Κοιτάξτε, σας συμβουλεύω να δείτε τον κανονισμό. Δέχεστε ερώτηση ή όχι. Εξακολουθώ να πιστεύω πως ως θέμα αρχή. είστε ο πρώτος πρόεδρος που δεν μας ε, ε, λέτε ποιος θέτει την ερώτηση. Άρα δεν δέχεστε την ερώτηση. Συνεχίζουμε λοιπόν, προχωράμε. Το λόγο έχει ο κύριο Σάκη για δύο λεπτά. Η κυρία Σάκη, με συγχωρείτε. Ευχαριστώ Πρόεδρε, Επίτροπε, συνάδελφε. Τα περιστατικά στο Ιράκ και στην όλη Μέση Ανατολή είναι πάρα πολύ ανησυχητικά, αλλά δεν προήλθε αυτό του. Το Ισλαμικό κράτος αναπτύχθηκε και με τις συνθήκες πολέμου στη Συρία, με την τοξική παρέμβαση κάποιων φορέων του Περσικού κόλπου και η Ισλαμική επιρροή στην πολιτική δεν αποτυπώνει τον πλουραλισμό που επικρατεί στη χώρα, στο Ιράκ. Η κατάσταση στο Ιράκ μετά τον πόλεμο ανέδειξε προβλήματα πολιτικής, οικονομικής φύσεως και αυτό οδήγησε στο εκρηκτικό σενάριο το οποίο αντιμετωπίζουμε σήμερα. Οι αξιώσεις, οι παράνομες αξιώσεις του χαλιφάτου, οι μαζικές εκτελέσεις, ο νόμος της Σαρίας αντιτίθενται στο διεθνέ ανθρωπίνο δίκαιο και θα πρέπει να λάβουν ένα τέρμα τώρα, αλλά να είμαστε και ρεαλιστέ σε ό,τι αφορά στο Ισλαμικό κράτο και να μην είμαστε δυσανάλογοι. Γιατί όλη η κατάσταση στην ε, Ιράκ χρειαζόμαστε μια πολιτική λύση και θα πρέπει να σεβόμαστε την επικυριαρχία του Ιράκ. Η έκκληση για την ανεξάρτηση για την εξαρτησία του κουρδικής ε, περιοχής είναι κατανοητή, αλλά ενδεχομένως να περιοδοτήσει περαιτέρω την κατάσταση που δεν θα ωφελήσει κανέναν σε αυτή τη φάση. Ξέρουμε ότι το IS έχει διάφορους Ευρωπαίους ε, ε, που μάχονται και αυτοί δεν θα πρέπει να, υπονομε... να υποτιμάται ο κίνδυνος όταν επιστρέψουν αυτοί οι άνθρωποι στις δικές μας ε, κοινωνίες. Θα χρειαστούμε λοιπόν μέτρα ασφάλειας για να αποτρέψουμε την διάδοση αυτών των ιδεολογιών που καλούν τον κόσμο να συμμετέχει στο τζιχάτ και επίσης θα πρέπει να συνεργαστούμε και με την Τουρκία μέσα από τις οποία πολλοί ε, επισέρχονται στο Ιράκ και στη Συρία και θα πρέπει να φροντίσουμε να υπάρξει μια βιώσιμη κατάσταση στη Μέση Ανατολή και προκειμένου να επιτύχουμε αυτό θα πρέπει να συμπεριλάβουμε και το Ιράν και στη Σαουδική Αραβία στις συζητήσεις γιατί και αυτοί έχουν πολλούς φορείς για να προσπίσουν τα επικίνδυνα συμφέροντά τους στην περιοχή. Σας ευχαριστώ. Υπάρχει μια ερώτηση για σας. Κυρία Σέικε, τη δέχεστε? Δέχεστε μια ερώτηση με μπλε κάρτα? Ναι, δεν σας ακούω. Εάν δεν πατήσετε το κουμπάκι δεν σας ακούω. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ. Ναι, δεν είχε ανάψει το μικρόφωνο μου. Ευχαρίστως να ακούσω ποιος είναι και να δεχτώ και την ερώτηση. Παρακαλώ κύριε Έτεριτς, την ερώτησή σας. Χαίρομαι που είχατε το θάρρος να δεχτείτε την ερώτηση. Θα με ενδιαφέρει πολύ να ακούσω τι έχετε να πείτε και αν συμφωνείτε μαζί μου ότι ο καλύτερο τρόπο να σταματήσουμε με τα περαιτέρω προβλήματα σε αυτή την περιοχή είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη τη να πάψουν να επεμβαίνουν με την εξωτερική του πολιτική που έχει ως αποτέλεσμα να καταστρέφονται άλλες χώρες, να μην στέλνει στρατεύματα πλέον πουθενά, εκτός εάν ε, υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη ανάγκη. I'm afraid, uh, dear... Λοιπόν, πολύ φοβάμαι, συνάδελφε, ότι τα πράγματα δεν είναι ασπρόμαυρα και δεν υπάρχει μια λύση που να ισχύει ενιαία για την Ευρώπη που θα πρέπει να διαδραματίσει το σημαντικό παγκόσμιο ρόλο τη προκειμένου να ανταπεξέλθει στι διάφορε προκλήσει. Είτε πρόκειται για παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, είτε για άλλε κρίσει. Όπω βλέπουμε στη Μέση Ανατολή, ιδιαίτερω τώρα, και πιστεύω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να αναλάβει πιο ηγετική θέση, να κάνει διπλωματικές προσπάθειες, να συνεργαστεί με τους εταίρους όπως την Τουρκία για να ανακάμψει τη διάδοση της βίας μέσω Τουρκίας σε χώρες όπως η Συρία και το Ιράκ. Υπάρχουν λοιπόν πολλά βήματα πριν από τη στρατιωτική παρέμβαση, αλλά όλοι ξέρουμε ότι δυστυχώς ο κόσμος ε, σε κάποιες περιπτώσεις ε, ζητάει και όχι μόνο ήπια μέσα, αλλά και σκληρά μέτρα. Ευχαριστώ. Ο κύριος Κόζο Περμούη, για 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αυτοί που είναι υπέρ τη ατιμορρησία ε, δεν είναι υπέρ της μνήμης. Εμείς έχουμε μνήμη όμως, ε, και ξέρουμε ότι η σημερινή κατάσταση στο Ιράκ δεν είναι φυσική καταστροφή. Έχει προηγούμενα. Και αυτές ήταν, αυτό ήταν σε σύνοδο στις Αζόρες που με κοροϊδία άνοιξε η πόρτα για την πρώτη γενοκτονία του 21ου αιώνα. 1,5 εκατομμύριο νεκροί ήδη ε, στο Ιράκ. Ο τότε πρόεδρος της Κομισιόν ε, Μπαρόσο ήταν ε, ο οικοδεσπότης αυτής της Συνόδου. Δεν πιστεύω ότι πρέπει να ξεχνάμε το διεθνές ε, δίκαιο. Δεν μπορούμε να αφήσουμε τους ε, τους εγκληματίες, γιατί η παρέμβασή τους, η κατοχή, είχε ως αποτέλεσμα να έχουμε σήμερα μια κατεστραμμένη, αποσταθεροποιημένη χώρα που είναι διαιρεμένη σε φυλές, σε εθνοτικές ομάδες και η σημερινή κυβέρνηση βλέπουμε να έχει τον εθνικό στρατό ε, ως πολιτοφυλακή ε, και να τους εξαπολύει αυτούς κατά των ε, διαδηλωτών, όπως το 2011 παραδείγματος χάρη. Επίσης βλέπουμε και τρομοκράτες, κάποιοι να στηρίζουν τη Συρία, κάποιοι τη Λιβύη και η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να ξεκινήσει μια νέα εξωτερική πολιτική, έχει αυτή τη δυνατότητα αν προωθήσει στο πλαίσιο του ΟΗΕ μια συνέλευση με τις αραβικές και γειτονικέ χώρες ώστε οι Ιρακινοί να έχουν πια ένα νέο σύνταγμα για όλους τους Ιρακινούς χωρίς εθνοτικά φιλετικά προβλήματα ώστε όλοι οι Ιρακινοί, όλες οι Ιρακινές να μπορούν να αποφασίσουν το μέλλον της χώρας τους και το μέλλον των φυσικών τους πόρων που επαναλαμβάνω και υπενθυμίζω σε αυτούς μόνο ανήκουν. Μόνο έτσι θα πετύχουμε την ειρήνη. Ευχαριστώ. Κύριε Κόζο Περμόη, δέχεστε την μπλε κάρτα. Ναι, δέχομαι. Η κυρία Αναγκόμα, παρακαλώ. Επειδή αναφερθήκατε στη μνήμη, το 2003 τα έχω καταδικάσει εγώ αυτά που έγιναν. Γιατί δεν πάτε πιο πίσω στην εποχή του Σαντάμ Χουσέιν ή θεωρείτε ότι ήταν δημοκράτης και όχι ένας φοβερός και τρομερός καταπιεστής δεν ευθύνεται και αυτός για αυτά που συμβαίνουν σήμερα, για τη βία, για τις φιλετικές ε, αυτές ε, ε, συγκρούσεις και όχι μόνο εντός και εκτός. Θέλετε να απαντήσετε παρακαλώ. Κοιτάξτε, το, το πρόβλημα είναι ότι έχετε επιλεκτική μνήμη, ξέρετε. Αυτό είναι το πρόβλημά σας. Εμένα πάει και στη μνήμη μου και πίσω στο βρετανικό υπεριαλισμό. Τα προβλήματα από τότε προέρχονται, από την απεικιοκρατία. Φυσικά αυτό που ε, συμβαίνει στο Ιράκ σήμερα οφείλεται στο 2003, αλλά και πιο πριν. Εγώ δεν έχω πρόβλημα. Θυμάμαι καλά ε, τον ε, Σαντάμ Χουσέιν. Ξέρετε, συγγενής μου, αδερφός μου συγκεκριμένα δολοφονήθηκε στο Ιράκ και πολλοί συμπατριώτες μου έχουν δολοφονηθεί. Δεν έχω εγώ πρόβλημα μνήμης. Σας ευχαριστώ. Το λόγο έχει ο κύριος Σμιθ για μισή λεπτά. Πρόεδρε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Όπω και πολλοί συνάδελφοι, έχω την αίσθηση ότι υπάρχει έντονα σύστηματα στη συζήτηση για το Ιράκ. Και εγώ θυμάμαι να περπατώ στο, στη και να διαμαρτύρομαι για την ε, παρέμβαση, την ε, εισβολή στο Ιράκ από την Συμμαχία των Προθήμων. Και από τότε, από αυτή την πράξη της τρέλας έχουν ε, περάσει έχουν περάσει χρόνια πολλά και σύμφωνα με εκτιμήσει του ΟΗΕ είναι μόνο στο Βόρειο Ιράκ 2,1 εκατομμύρια των εσωτερικά εκτοπισμένων. Είναι πάρα πολύ περίπλοκη λοιπόν η κατάσταση. Ο ρόλο μα ω Ευρωπαϊκή Ένωση, πέρα από το να θυμόμαστε το πώ φτάσαμε εδώ που φτάσαμε και δεν θα πρέπει να υπάρχει τίποτα που να το ξεχνάμε. Πέρα από αυτό όμως θα πρέπει να βρούμε το δρόμο για να βγούμε από τον εφιάλτη αυτό. Και θα ήθελα να αναφερθώ σε τρία θέματα στη συζήτηση αυτή. Το ρόλο των Κούρδων, το ρόλο του Ιράν, το ρόλο τη Ασαντική Αραβία στον Περσικό κόλπο. Αν και υποστηρίζω το υπόλοιπο ψήφισμα, το οποίο πραγματικά είναι αξιέπαινο και θεωρώ ότι έχει το σωστό πνεύμα. Σε ό,τι αφορά το ρόλο των Κούρδων στο ΕΕΦ, σημειώνουμε τον ρόλο της κουρδικής ε, κυβέρνησης, περιφερειακής κυβέρνησης, σε ό,τι αφορά τις ε, επιπρόσθετες ε, περιοχές και ασκούμε κριτική στις δράσεις αυτές, θεωρώ ότι αυτό είναι ρεαλιστικό και πραγματιστικό. Στο, στην αιτηλογική σκέψη G αναφέρουμε πόσο τι ισχύει για θέματα τζιχάτ και το βάρος που επιφορτίζει πολλούς ε, πρόσφυγες. Αλλά στο σημείο 11 αναφέρουμε ότι οποιαδήποτε συνταγματική αλλαγή θα πρέπει να σέβεται μία σωστή διαδικασία σε ό,τι αφορά τα δικαιώματα των μη κουρδικών μειονοτήτων που ζουν στην περιφέρεια. Και αυτό θα πρέπει να το προωθήσουμε. Σε ό,τι αφορά το ρόλο του Ιράν στο σημείο 9, καλούμε και αυτό είναι σημαντικό την εθνική, την εθνική κοινότητα και κυρίω εμά να διευκολύνει τον περιφερειακό διάλογο σε ό,τι αφορά τα προβλήματα τη Μέση Ανατολή και να συμπεριληφθούν οι σημαντικοί παράγοντε και ότι οι όμορε χώρε του Ιράκ δεν μπορούν να θα θεωρηθούν άσχετες και θα πρέπει να συμμετέχουν και αυτές στην εξέβρεση της λύσης. Πρόεδρε, δεν μπορούμε να αρνηθούμε το ρόλο μας στη δημιουργία της κατάστασης στο Ιράκ. Δεν μπορούμε λοιπόν να αποφύγουμε παρά να βρούμε έναν τρόπο να βγούμε από τον εφιάλτη. Σας ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος James Carver για τρία λεπτά. Κύριε Πρόεδρε, το Ιράκ έχει να καταδείξει την αποτυχία των δυτικών κρατών. Αυτό αποτελεί ένα σκάνδαλο. Έχουν αποτύχει, λοιπόν, έχουμε αποτύχει και πριν από 100 χρόνια είχαμε αποτύχει σε ό,τι αφορά τις ε, διαφορές αυτές, τις άλλαγες αυτές. Ο Ιρακινός λαός και πιστεύω ότι ο δεύτερος Περσικός πόλεμος προετοίμασε όχι τη νίκη, αλλά όχι τη ζωή μετά τη νίκη. Και ναι, οι μπαθιστές έπρεπε να αφαιρεθούν από το Ιράκ, αλλά αυτό που ακολούθησε ήταν η μεγαλύτερη αποτυχία της σύγχρονης εποχής σε ό,τι αφορά την εξωτερική πολιτική. Η καταστροφή του στρατιωτικού σκέλους του Ιράκ μετά την πτώση του Σαντάμ και Αντιμετωπίζουμε λοιπόν ένα τεράστιο πλωστάσιο το οποίο ουσιαστικά εγκαταλείφθηκε και αυτό οδήγησε σε αιματηρές συγκρούσεις στα πλαίσια της, ε, του ίσης τώρα. Και τώρα λοιπόν έχουμε πετύχει ακριβώς το αντίθετο. Ο Αλμαλακή έχει αποδειχθεί εντελώς ακατάλληλος ε, για τη δουλειά του και αυτό υπογραμμίζει την ε, ανευθυνότητα των δυτικών ηγετών και ο Αλμαλίκη αγνοεί τους Κούρδους και τους Σουνίτες στην περιοχή. Άρα ο κόσμος τώρα μόνο να προσευχηθεί μπορεί και οι Βρετανικές εφημερίδες αναφέρουν ότι περίπου 15.000 Βρετανοί μουσουλμάνοι έχουν ταχθεί στο πλευρό της ίσης. Και έτσι έχουν εισέλθει στην Ήπειρό μας και υποσκάπτουν τρομοκρατικές εκστρατείες. Πέρσι λοιπόν αποφύχθη η συλλογή τέτοιων στοιχείων δεδομένων στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τους ταξιδιώτες. Οι ίσες έχουν κλέψει 400 εκατομμύρια ευρώ από τράπεζες και έτσι είναι μία από τις χειρότερες ε, τρομοκρατικές οργανώσεις. Θα μπορούσαν να αποσταθεροποιήσουν την περιοχή και όλο τον κόσμο κατά συνέπεια. Θα πρέπει λοιπόν αυτό να αποτελέσει ένα μήνυμα για μα, Όταν θα πρέπει να λαμβάνονται αποφάσεις, θα πρέπει να λαμβάνονται όσο γίνεται με μεγαλύτερη ενημέρωση από τη Μέση Ανατολή, από τον ΟΗΕ και με την αρμοδιότητα του ΟΗΕ. Η Βρετανία λοιπόν μπήκε στον πόλεμο αυτό με τον Ιράκ λόγω της ε, ε, περίεργης του Τόνι Μπλερ. 179 Βρετανοί, γενναίοι Βρετανοί, έχουν θυσιαστεί και πολλοί, πολλοί άλλοι έχουν υποστεί ψυχολογικά δράματα ή σωματικά, ε, σωματικές ε, τραυματισμούς, ε, τους οποίους θα πρέπει να αντέξουν και να υποφέρουν την υπόλοιπη ζωή τους. Δεν θέλουμε λοιπόν άλλο βρετανικό αίμα να χυθεί. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ. Και τώρα ο κύριος Μάριο Μποργέτσιο για δύο λεπτά. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Εντυπωσιακή ταχύτητα με την οποία αυτή σε δυνάμεις 15.000 ανδρών έχει κατακτήσει ένα μέγα μέρος του Ιράκ θα πρέπει να μας κάνει να ανησυχήσουμε και για αυτή την κατάσταση που χτυπάει την πόρτα του, της Ευρώπης. Σίγουρα πρόκειται για πλήρη αποτυχία της ε, ε πολιτικής του Ομπάμα για την τρομοκρατία που ασχολήθηκε αποκλειστικά με την Αλκάιντα και αγνόησε τις τεράστιες δυνατότητες που μπορεί να έχει ο Ισλαμικός εξτρεμισμός σε μια ολόκληρη σειρά από οργανώσεις που είναι δύσκολο είναι να ελέγξει κανείς και εντός των οποίων λειτουργούν και 2-3 χιλιάδες μαχητές του Αλάχ που έχουν γεννηθεί και κατοικούν την Ευρώπη μας και που πιθανότατα θα επιστρέψουν σπίτια τους, θα ζήσουν ανάμεσά μας. Θα τους ξαναδούμε και ίσως θα τους ξαναβρούμε ανάμεσά μας έτοιμους να δράσουν με τον τρόπο που είδαμε. Και αυτό θα πρέπει να μας κάνει να τρέμε τρέμομαι, να τρέμουμε εδώ στην Ευρώπη που ωστόσο στις απαντήσεις της δείχνει να είναι αυτή η οποία σωστά την έχει περιγράψει η σπουδαία ε, συγγραφέα Σοριάννα Φαλάτσι της Ιταλίας. Δεν μπορούμε να ε, παραβλέψουμε άλλωστε τον ε, βία ομιλία του μαύρου χαλίφη της Βαγδάτης που λέει ότι πολύ περισσότερα αφορά όλους τους μουσουλμάνους αυτή ο πόλεμος τους οποίους ζητά να συμβάλλουν δραστήρια στο τζιχάντ, στον Ιερό Πόλεμο και μάλιστα και στην κατάκριση της Ρώμης που θεωρείται ο γεωπολιτικός στόχος καθώς είναι το κέντρο της του χριστιανισμού και των και ο κληρονόμος ε, των σταυροφοριών. Η Ευρώπη μόνο αν είναι τυφλή μπορεί να κάνει πως δεν καταλαβαίνει. Πρόκειται για εξτρεμισμό που δεν θέτει πλέον σύνορα εδαφικά. Αφορά ολόκληρο τον κόσμο τον τζιχάντα αυτό και η Ευρώπη μας ε, θεωρείται ως ε, έδαφος η προσκατάκτηση. Πώς μπορούμε να μην καταλαβαίνουμε ότι έχουμε μπροστά μας τέτοιου είδους πρόκληση. Σας ευχαριστώ. Το λόγο έχει ο κύριος Κέλαμε για δύο λεπτά. Παρακαλώ. Σας ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Το Ιράκ αντιμετωπίζει υπαρξιακή κρίση και η κυριότητά του διακυβεύεται αυτή τη στιγμή. Το θέμα είναι πώς ήταν δυνατόν κάποιες ομάδες τρομοκρατών μπόρεσαν να πάρουν τον έλεγχο τόσο μεγάλων μερών ε, κομματιών αυτής της χώρας μέσα σε λίγες εβδομάδες. Νομίζω πως την ευθύνη έχει και η Ιρακινή κυβέρνηση, η οποία τα τελευταία δέκα χρόνια η, η κυβέρνηση Αλμαλίκη απέτυχε να ηγηθεί ενός συνασπισμού που θα αγκάλιαζε όλους τους τομείς της, ευρωπαϊκής, της Ιρακινής πραγματικότητας. Αντίθετα, περιθωριοποίησε την κοινότητα των Σουνιτών, τους Κούρδους, τους αρνήθηκε τη συμμετοχή και εξαρτόταν διαρκώς και όλο και περισσότερο από την στήριξη του Ιράν. Ως αποτέλεσμα, η κυβέρνηση Αλμαλίκη ε, σαφώς αποδυνάμωσε τη στήριξή της, την υποστήριξη που είχε μάλλον από τη χώρα και ε, τα κίνητρα για να, και έδωσε κίνητρα για να στηριχθούν οι τρομοκράτες. Χρειαζόμαστε μια νέα κυβέρνηση εθνική εμφυλίωσης που θα τίνει χείρα μετριοπάθεια στους μετριοπαθείς Σουνίτες και, και στους ηγέτες των Κούρδων. Οι, Ευρωπαϊκοί, οι Ευρωπαίοι ηγέτε θα πρέπει να πιέσουν όλε τι μετριοπαθεί δυνάμει ώστε να επιτευχθεί συνένεση. Καλούμε επίση την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να στείλει περισσότερη ανθρωπιστική βοήθεια από την πρόσφατη αύξηση των 12 εκατομμυρίων γιατί υπάρχουν σχεδόν 2 εκατομμύρια εσωτερικά εκτοπισμένα άτομα. Πρόσφατα πολλά εκατομμύρια έφυγαν από τη Μοσούλη και χρειάζονται άμεση στέγαση και ιατρική περίθαλψη. Οι Κούρδοι που χρειάστηκαν να δεχτούν το μεγαλύτερο μέρος αυτών των προσφύγων χρειάζονται και αυτή η βοήθεια. Και τέλος ανησυχώ πάρα πολύ για το μέλλον των χριστιανικών κοινοτήτων του Ιράκ, των οποίων τα νούμερα μειώθηκαν κατά δύο τρίτα τα τελευταία εννέα χρόνια. Στο Ιράκ πάνω από 300.000 αφέθηκαν να αντιμετωπίζουν διαρκή παρενόχληση και διώξεις. Οι χριστιανοί μάλιστα είναι αυτοί που δεν καταφεύγουν στη βία και είναι ζωτική σημασία για την καθίδρυση διαλόγου και για τη γεφύρωση των κενών. Δίνουν, παρέχουν ε, τη βάση για την παιδεία σε ολόκληρη την περιφέρεια. Μάλιστα ασκούν ένα ρόλο ένταξης και αλληλεγγύης μια, σε μια αποσυντηθέμενη κοινωνία. Είναι ρόλος μας να τους βοηθήσουμε. Σας ευχαριστώ κύριε Κέλα. Υπάρχει ε, μπλε κάρτα για εσάς. Τη δέχεστε. Δέχεστε μια ερώτηση. Μπλε κάρτα που σας απευθύνεται. Πολύ ωραία. Οπότε το λόγο έχει ο Ντουάρ Φερό. 30 δευτερόλεπτα άνευ μικροφώνου. Σας ευχαριστώ για την παρέμβασή σας. Πράγματι δεν υπάρχουν μόνο οι Σουνίτες και οι στο Ιράκ, υπάρχουν και χριστιανοί. Χριστιανοί λησμονημένοι. Σήμερα οι χριστιανοί μπορούν να επιλέξουν είτε το να φύγουν είτε το να εκτελεστούν. Σήμερα οι χριστιανοί, κύριοι, ε, και είναι απλό το ερώτημά μου, έχουν το δικαίωμα οι χριστιανοί σήμερα ακόμη να κατοικούν ε, στην Εγγύης Ανατολή, ναι ή όχι. Σας ευχαριστώ πολύ για αυτό το ερώτημα. Είναι και δικό μου ερώτημα και δική μου απορία όμως. Νομίζω ότι είναι κοινή απορία και των δυο μας. Ε, η κατάσταση, η μοίρα των χριστιανών στην στην Ανατολή δυστυχώ φαίνεται να έχει αποφασιστεί. Ο κύριος Χόιτο έχει το λόγο για τρία λεπτά. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Καταρχάς θα ήθελα να εκφράσω τη βαθιά μου ανησυχία για την κλιμάκωση της βίας και την επιδείνωση της κατάστασης στο Ιράκ με βάση ε, τα Ηνωμένα Έθνη 1,2 εκατομμύρια είναι εσωτερικοί εντοπιστέντες ε, εντός ε, του Βόρειου Ιράκ και θα πρέπει να χαιρετήσουμε τα επιπλέον 7 εκατομμύρια ευρώ που δίνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για Ανθρωπιστική Βοήθεια ακούμε ε, αφρικιαστικές ε, καταστάσεις ε, για τη δολοφονία ενός 18χρονου και ενός 44χρονου από τους μαχητές του Ισλαμικού κράτους. Πραγματικά Βιοπραγίες είναι καθημερινό φαινόμενο σε βάρος αμάχων. Ζητούμε το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου από όλες τις πλευρές. Η ε, Human Rights Watch έκανε στις 11 Ιουλίου, ε, μάλλον δημοσίευσε μία έρευνα. Φαίνεται να υπάρχουν 255 παράνομες εκτελέσεις ε, κρατουμένων για αντίπεινα. Πρέπει να σταματήσουν όλα αυτά. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να μιλάει για συμφωνίες. Πώς θα προωθήσουμε τα ανθρώπινα δικαιώματα, το κράτος δικαίου εάν δεν αντιμετωπίσουμε τις πάρα πολύ σοβαρές αυτές απειλές που υπάρχουν, ιδίω από τα κράτη παρή στην περιοχή. Δεν μπορούμε να ε, δαπανίσουμε άλλο χρόνο για να συζητάμε τις αιτίε. Η σουνητική ε, μειοψηφία στο Ιράκ δεν εκπροσωπείται. Ο Μακ Τσαμπούρη ορίστηκε πρόεδρος του Κοινοβουλίου στο Ιράκ και ελπίζουμε να βοηθήσει στην αποκλιμάκωση της κατάστασης και σίγουρα πρέπει να δούμε και τι γίνεται με την ένταση μεταξύ Βαγδάτη και ε, Αρμπίλ. Το Κουρδιστάν, λέει ο Μαλίκη, είναι ένα καταφύγιο για τους ε, τρομοκράτες. Δεν βοηθούν τέτοιες ε, δηλώσεις. Πολλοί είναι αυτοί οι οποίοι έχουν φύγει προς το Κουρδιστάν για να γλιτώσουν αλλά η πρόσβαση και η είσοδος έχει περιοριστεί. Ε, παρότι υπάρχουν πάρα πολλοί οποίοι προσπαθούν να, φύγουν, να διαφύγουν από τη βία. Τα κουρδικά πολιτικά ε, δικαιώματα πρέπει να αναγνωριστούν και πρέπει να υπάρξει διάλογος μεταξύ Κούρδων και Ιρακινών. Καταστροφή ήταν η καθυστέρηση σχηματισμού κυβέρνησης από τον Αλμαλίκη και μεγάλος κίνδυνος για το μέλλον του Ιράκ. Τώρα θα πρέπει η Ιρακινή κυβέρνηση να εστιάσει στην εθνική ενότητα. Γι' αυτό καλούμε όλους του πολιτικού ηγέτες, ιδίω τον Πρωθυπουργό, να φροντίσουν να υπάρξει μια κυβέρνηση αλληλεγγύη που θα εκπροσωπεί ε, την πολυμορφία ε, του Ιρακινού πληθυσμού. Επίσης ε, έχουμε μία σχέση μεταξύ της ανόδου του Ίσης ε, και του εμφύλιου στη Συρία και αυτό θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε συνολικά το πρόβλημα ε, το μεσανατολικό. Διακόπτεται ο μιλητής. Ευχαριστώ πολύ. 1,5 λεπτό τώρα έχει το λόγο ο κύριος Μπέλντερ. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Είναι εντυπωσιακό, το, εντυπωσιακό ότι στο ψήφισμα αυτό δεν αναφέρεται κανένας ε, λόγος για τον ρόλο της Τουρκίας στις ε, θυελώδες εξέλιξεις στο Ιράκ και θα ήθελα να ακούσω μία απάντηση από το Συμβούλιο σε ό,τι αφορά το θέμα αυτό για τη σοβαρή αιτίαση ότι η Τουρκία έχει συγγραμματοποτήσει το χαλιφάτο της ε, ίσης με την αγορά πετρελαίου. Είναι πολύ σοβαρό αυτό σε ό,τι αφορά και την κατάκτηση του μεγαλύτερου οπλοστασίου του Ιράκ από πλευρά τη ΙΣΙΣ. Και από το Κουρδιστάν εκτοκτεύονται κατηγορίες σήμερα ότι η ΙΣΙΣ και το χημικό της οπλοστάσιο χρησιμοποιείται κατά των Κούρδων. Το Συμβούλιο γνωρίζει αυτές τις ανησυχητικές ειδήσει και πώς αξιολογεί την κατάσταση. Σίγουρα οι εκθέσεις αυτές για το χημικό πλωστάσιο στην Αμουταρά ε, με τις πυράβλους με το αέριο Σαρίν είναι πάρα πολύ Έχουν γίνει συζητήσει μεταξύ Βρυξελών και Βαγδάτης και θα θέλαμε λοιπόν να δοθεί ιδιαίτερη σημασία στην δραματικά μειωμένη χριστιανική μειονότητα στο Ιράκ και θα θέλαμε λοιπόν να ταχθούμε υπέρ της ε, παρουσίας και στο μέλλον των χριστιανών στη Μεσοποταμία. Θα θέλα λοιπόν να ε, γίνουν ψηφίσματα, αλλά δεν θέλουμε λόγια, θέλουμε δράσεις. Ευχαριστώ πολύ ο κύριος Νάρτ για 1,5 λεπτό. πρέπει να διερωτηθούμε πώς το ίσις κατάφερε μέσα σε λίγες μέρες ε, σχεδόν το μισό Ιράκ ε, να το καταστήσει και θα πρέπει να δούμε πώς οι Ταλιμπάν μπόρεσαν πάρα πολύ εύκολα τους Μουτσαχεντίν να τους εξολοθρεύσουν. Αυτό σημαίνει η υποστήριξη ε, του πληθυσμού είναι αυτό που βοηθάει μας αρέσει είτε όχι. Έχουμε μια σεκταριστική κυβέρνηση, την κυβέρνηση του Νούρι Αλ Μαλίκη. Ε, ε, όταν αναφερνόταν στην Νικαράγουα είχε πει ότι ναι αναγνωρίζω ότι είναι μπάσταρδος αυτός, αλλά είναι δικός μας μπάσταρδος. Ε, επομένως, έχουμε και αυτό το κίνδυνο ε, της βαλκανοποίησης ε, που μπορεί το Ιράκ να το κάνει ένα πραγματικό λαβέρνηθο για όλη τη Μέση Ανατολή. Δεν θα πρέπει να κοιτάμε προς το παρελθόν και τις περασμένες αμαρτίες, αλλά να κοιτάμε το μέλλον και να απαιτήσουμε να μην μιλάμε για δημοκρατικές ε, ε, εκλογές στο Ιράκ. Είναι πραγματικά ε, αντίφαση εξορισμού αυτό και είναι με μια φενάκι. Δεν μπορεί να συμβεί. Αλλά ας ζητήσουμε τουλάχιστον αλλαγή πλεύση από την κυβέρνηση Νόρια Αλμαλίκη. Ο κύριος Γκολνής για δύο λεπτά. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Επειδή Υπάρχουν, ε, έχουν περάσει 40 χρόνια από την ε, Ινδοκίνα. Ζούμε την απόρρεια της ε, εξαιρετικής πολιτικής ε, των Αμερικανών αυτή τη στιγμή στη Μέση Ανατολή. Και φυσικά με επικρία και ηρωνικά τα λέω αυτό. Αυτή η πολιτική στη Μέση και στην Αγγής Ανατολή στην ουσία ε, σημαίνει μεθοδική και άγρια καταστροφή της μόνης πολιτικής δύναμης που ήταν σε θέση να αντισταθεί στο πιο ριζοσπαστικό και το πιο κατακτητικό Ισλαμισμό, δηλαδή τον αραβικό εθνικισμό. Ο καθένας θα έπρεπε να έχει στο μυαλό του τα κρατικά ψέματα όπως ε, την υποτιθέμενη συμμετοχή του Ιράκ στις ε, επιθέσεις της 11 Σεπτεμβρίου που το Ιράκ δεν είχε καμία ευθύνη όπως τα υποτιθέμενα μέσα μαζικής καταστροφής. Ο κ. Δανοζάν είπε πως, σωστά πως δεν αρκεί η μνήμη αλλά χρησιμεύει πάντως για να μην κάνουμε ξανά τα ίδια λάθη και να μην πω και τα ίδια εγκλήματα. Θυμάστε τον κύριο Μπούς και τον κύριο Κόλιν Πάουελ που στο ΝΟΙΕ μέσα στη συνέλευση κουνούσε έτσι με βία αυτή το φιαλί που υποτίθεται είχε επικίνδυνα χημικά, χημικές ουσίες εκεί μέσα, ενώ είχε μόνο χρωματιστό νερό. Όλοι θα θυμάστε την ε, πραγματικά φρικαλέα ε, θανάτωση του Σαντάμ Χουσέιν, που δεν ήταν κανένα δημοκράτης βεβαίως, αλλά σίγουρα προστάτευε τις μειονότητες, όπως τη χριστιανική που αυτή τη στιγμή είναι είδος προ εξαφάνιση. Ε, αυτή τη στιγμή βλέπουμε τις Σουνίτες, Σουίτες και μια, την ανάδυση μιας ακόμα χειρότερης και πιο δυνατής δύναμης. Μερικές χιλιάδες ε, ε, μαχητές έχει τον Ιρακινό στρατό που υποτίθεται τόσο καταπληκτικά είχαν εκπαιδεύσει οι Αμερικανοί τον τσάκισε. Και τι κάνει, βασίζεται στους Σιήτες και στους Ιρανούς. Πρέπει να ολοκληρώσετε, κύριε Γκόλνης. Οι Αμερικανοί δεν θέλουν να συζητήσουν ακόμα με τους Ιρανούς. Ε, πραγματικά είναι μια καταστροφική πολιτική. Eh, κύριε Ντελάγκα, ευχαριστώ πάρα πολύ, Πρόεδρε. Με ντροπή διαπιστώνω ότι μια... χρειάστηκε μια επίθεση σε εμά, το δικό μας ε, σπίτι, για να καταλάβουμε τι συμβαίνει στο Ιράκ. Έγινε η επίθεση στις Βρυξέλλες στο Εβραϊκό Μουσείο και ε, καταλαβαίνουμε λοιπόν τι γίνεται στο Ιράκ. Αναφέρθηκε ότι η διεθνή κοινότητα ήταν ε, έκπληκτη από την επίθεση αυτή. Δεν συμφωνώ. Ε, δεν συμφωνώ. Είδαμε τι έγινε τα τελευταία δέκα χρόνια με την εκδίωξη σημαντικών ε, τμήματων του πληθυσμού στο Ιράκ, ε, ρεζοσπαστικοποίηση. Δεν μπορεί να ισχυριζόμαστε ότι ήταν ε, έκπληξη, αλλά ήταν μάλλον απαραίτητη η επίθεση στη Βρυξέλλε για να ξυπνήσουμε. Η πρώτη λοιπόν αντίδραση θα πρέπει να είναι η αντίδραση της ανθρωπιστικής βοήθειας. Και θεωρώ ότι τα 5 εκατομμύρια ε, επιπλέον τα οποία ε, αναφέρονται είναι σημαντικά. Κατά δεύτερον, ως Ευρώπη θα πρέπει να εξετάσουμε τις συνέπειες σε ό,τι αφορά την ασφάλεια της σπαστικοποίησης στο, στη Συρία, στο Ιράκ και θα πρέπει να προσπαθήσουμε να περιορίσουμε τις συνέπειες αυτές. Την προηγούμενη εβδομάδα έγιναν τέτοιες συζητήσει, αλλά είναι όλα μη δεσμευτικά. Η Ευρωπόλε αναφέρει και ότι χαρτογραφεί τους τρομοκράτες στην Ευρώπη και αυτό το μητρό δεν θα πρέπει να είναι κάτι ε, προαιρετικό, θα πρέπει να είναι υποχρεωτικό και κατά τρίτον θα πρέπει να υποστηρίξουμε τις ε, ε, μετριοπαθείς δυνάμεις στη χώρα αυτή. θα πρέπει να κοιτάξουμε τις ε, μετριοπαθείς ε, θρησκευτικέ κοινότητες. Ε, οι χριστιανοί, για παράδειγμα, που δεν θέλουν να διασπαστεί η χώρα, που έχουν σχολεία, που έχουν νοσοκομεία. Πρόκειται για μέρη όπου συνενώνονται ο κόσμος. Αν θέλουμε λοιπόν να έχει κάποια ευκαιρία για το μέλλον η χώρα αυτή, θα πρέπει να βοηθήσουμε και να προωθήσουμε την ανάπτυξη. Στην Βόρεια Ιρλανδία λοιπόν η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δράσει έτσι. Σας παρακαλώ λοιπόν να κάνουμε το ίδιο και στο Ιράκ. Ζήλ Παρνιό, ένα λεπτό. Ευχαριστώ Αγαπητοί Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, είναι κατεπήγον να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα στο Ιράκ. Βία, μυσαλλοδοξία, θρησκευτική ανελευθερία. Αυτό στο 55% του εδάφους του Ιράκ με τη δημιουργία του αυτού του Ισλαμικού κράτους θα πρέπει σίγουρα να στήριξουμε ανθρωπιστικά και οικονομικά το Ιράκ, όμως ταυτόχρονα θα πρέπει να επιδείξουμε πολιτικό σθένος. Χρειάζεται διπλωματική πολιτική εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα είναι ξεκάθαρη. Αυτό το σθένος το πολιτικό θα πρέπει να μας επιτρέψει να πούμε και ελπίζω να γραφεί και στο ψήφισμά μας ότι πρέπει κατεπηγόντως ε, να βρούμε πολιτική λύση για να υπάρξει κυβέρνηση εθνικής ενότητας αλλά χωρίς τον σημερινό Πρωθυπουργό. Μόνο αυτό θα μπορούσε να εξασφαλίσει την εδαφική ακαιρεότητα της χώρας. Είναι πολύ σημαντικό να συμπεριληφθεί το σημείο αυτό στο ψήφισμά μας ε, διότι αλλιώς ε, θα δημιουργήσουμε ε, ένα ακόμα μεγαλύτερο χάσμα μεταξύ Σουνιτών Σιητών. Ο κύριος Βανόρντιν έχει τώρα το λόγο για ένα λεπτό έχει κανένα νόημα εμείς οι βουλευτές, καταρχάς ε, είναι το ερώτημά μου, να συζητάμε το θέμα αυτό όταν δεν υπάρχει κάτι καινούριο ε, για να συζητήσουμε τελικά. Το γεγονός είναι ότι οι βουλευτές εδώ λίγο μπορούμε να επηρεάσουμε την κατάσταση. Η Κομισιόν δεν κατέληψε την αίθουσα. αλλά βάζουν το χέρι τους ε, ε, στην ανθρωπιστική βοήθεια, στα χρήματα δηλαδή. Αυτοί τα ελέγχουν. Οι ε, τη Κομισιόν όμως απέχουν από αυτή τη συζήτηση. Η Συρία φλέγεται, η Χαμάς σφίγγει και αυτή τις γροθιές της στο, στην Παλαιστίνη. Γνωρίζουμε τα, τα προγράμματα εξοπλισμού, πυράβλων, στη Μέση Ανατολή. Σίγουρα πρέπει να αλλάξει κατάσταση στο Ιράκ. Έχουμε δαπανίσει πάρα πολλά χρήματα. Ένα δις έδωσε η Ευρωπαϊκή Ένωση για το Ιράκ. Αλλά το ένα τέταρτο του πληθυσμού ζει με 2 δολάρια ή λιγότερο την ημέρα. Η υδροδότηση, η αποχέτευση, ε, έχουν καταστραφεί τα συστήματα αυτά. Παρά τεράστιες ε, δαπάνες από πλευράς της διεθνούς κοινότητας και βλέπουμε πλέον να αναδύεται και ένα νέο τρομοκρατικό κράτος. Με αυτό το στρατό του Ίσης, ε, το στρατό των δολοφόνων που απειλεί την ε, Βαγδάτη. Τελευταία διεθνής διάσκεψη για το Ιράκ έλαβε χώρα το 2003. Πρέπει να ολοκληρώσετε, λέει η Δεν πιστεύω ότι είναι καιρό ο ΙΕ να συγκαλέσει μια νέα διάσκεψη για να βοηθήσουμε ε, να υπάρξει μια σταθεροποίηση στο Ιράκ και πρέπει να δούμε πιο προσεκτικά πώς δαπανώνται οι πόροι μας. Πού δαπανώνται οι πόροι μας. Ευχαριστώ. Πρόεδρος. Κυρία Μπιλμπάου Μπαραντίκα για 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Στο Ιράκ καταρχάς υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα κοινωνικής αδικίας και ε, ανελευθερίας που πλήττει του περισσότερου Ιρακινού, είναι ένα εργοστάσιο που παράγει απόγνωση σήμερα το Ιράκ και καλλιεργεί και υποθάλπει εξτρεμισμού. Είναι μεγάλα τα στρατηγικά ε, συμφέροντα και δυστυχώς ε, έχει γίνει ένα ε, μια πυρητιδαποθήκη θα έλεγα η περιοχή αυτή. Δεν είναι μόνο θέμα ασφάλειας, στρατιωτικό το θέμα, πολύ περισσότερα διακυβεύονται. Θα πρέπει να βρούμε τη ρίζα του προβλήματος ε, και να, και να επιλύσουμε το θέμα. Υπάρχουν ανισότητες, καταπίεση, δεν ε, γίνονται σεβαστά τα θεμελιώδη δικαιώματα. Η ακαιρεότητα επίσης ε, του κράτους. Όταν δεν δίνει απαντήσεις ε, το κράτος στα προβλήματα των πολιτών, όλα τα λένε ένα λόγια. Γι' αυτό θα πρέπει να στηρίξουμε μια ολοκληρωμένη πολιτική, κοινωνική και οικονομική λύση για το πρόβλημα του Ιράκ. Στηρίζω ε, την αναγγελία της κυβέρνησης του Κουρδιστάν να κάνει δημοψήφισμα για τις μειονότητες. Οι πέντε ομάδες αυτό λένε στο ε, ψήφισμά τους. Ελπίζω να ε, σχηματιστεί μια σταθερή κυβέρνηση σύντομα με βάση τον περιφερειακό διάλογο. Στο μεταξύ πάντως πρέπει να στηρίζουμε με διπλωματική και ανθρωπιστική βοήθεια το Ιράκ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Γκρζίπ. Για δύο λεπτά. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η κατάσταση εξακολουθεί να είναι σοβαρά το δει. Γιατί το Ισλαμικό κράτος ε, αποτελεί το στόχο όλων των μαχητών. Πέρα από όλα αυτά, υπάρχει μεγάλα παραβίαση των, των ανθρώπινων δικαιωμάτων. Η ανθρωπιστική κατάσταση είναι επίσης πάρα πολύ ανησυχητική και θα πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερη σημασία στην κατάσταση αυτή, γιατί το Φεβρουάριο την τελευταία φορά που συζητήσαμε εδώ στο Κοινοβούλιο την κατάσταση στο Ιράκ, αντέφερα την επιδείνωση της ιστορικής κατάστασης στο Ιράκ και ιδιαίτερος σε ό,τι αφορά τις χριστιανικές μειονότητες και σε ό,τι αφορά όλα τα εκτοπιστάντα άτομα. Έκτοτε η κατάσταση έχει επιδεινωθεί περαιτέρω. Οι σχέσεις δε μεταξύ της ε, κεντρικής κυβέρνησης και της κουρδικής μειονότητας έχει τεθεί υπό και ενδεχομένως να αντιμετωπίσουμε ένα τελείως ε, νέο κράτος ε, των Ιρακινών Κούρδων. Αυτό να το επιθυμούμε. Και ίσως αυτά τα αιτήματα για τον κουρδικό κράτος να είναι κάτι το λανθασμένο σε ό,τι αφορά και τα δικαιώματα των Συνητών, των ζητών και των Κούρδων. Επίσης, βλέπουμε ότι είναι δυσανάλογα μεγάλος ο αριθμό των εκτοπιστέντων και στις δύο κοινότητε. και υπάρχει μεγάλη απειλή ανοιχτή ε, σύραξης. Αυτό το έχει επισημάνει και ο Ιρακινός ε, χριστιανός ε, επίσκοπος που θα ήθελε να οικοδομηθούν γέφυρες μεταξύ των δύο αυτών κοινοτήτων προκειμένου να αποφευχθεί ενδεχόμενη ανθρωπιστική κρίση, γενοκτονία. Πραγματικά είναι μεγάλη απειλή. Ένα λεπτό, ο κύριος Ζεμκέ. Σας ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Η συζήτηση που κάνουμε σήμερα αφορά ναι, το Ιράκ που βρίσκεται στο χείλος της εξαφάνισης γιατί από τη πλευρά βλέπουμε το, την ανάδυση του χαλιφάτου των Σουνιτών και από την άλλη ένα νέο κουρδικό κράτος. Παρά όλα αυτά είμαι της άποψης ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα πρέπει να αναμειχθεί με στατητικό τρόπο για να στηρίξει οποιαδήποτε από αυτές τις πλευρές ε, στο πλαίσιο αυτού, αυτής της ε, σύγκρουσης. Αυτό που θα πρέπει να κάνουμε είναι να ασκήσουμε πίεση στη νέα Ιρακινή κυβέρνηση ώστε να δημιουργήσει νέες δομές, νέες δομές που θα λάβουν υπόψη τα συμφέροντα των μειονοτήτων των ΣΥΤΟΝ και των Σουνιτών και έτσι να προκύψει μια ειρηνική λύση σε αυτή την κατάσταση. Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, το βασικό πρόβλημα είναι ο Πρωθυπουργό Αλμαλίκη που ενεργεί ω δικτάτορα. Έχει προκαλέσει τη σημερινή κρίση λόγω των ε, ε, κατασταλτικών του πολιτικών κατά των ε, του λαού των Ιρακινών επίσης κατά των Κούρδων. Η λύση είναι να απομακρυνθεί ο Αλμαλίκη που είναι ε, μαριονέτα του Ιρανικού καθεστώτος. Ε, θα πρέπει να σταματήσουμε την παρέμβαση, την επέμβαση μάλλον του Ιρανικού καθεστώτος γιατί αυτό είναι, αυτή είναι το βασικό πρόβλημα για ολόκληρη την περιοχή. Οι νεαροί Σουνίτες και οι ξένοι στερετικοί ε, αυτό μας έχουν πει. Πρέπει να στηρίξουμε το αίτημα του Ιρακινού λαού για αλλαγή και για μια πραγματική κυβέρνηση για όλους. Αν δεν απομακρυνθεί ο Αλμαλίκη ε, θα υπάρξει όλο ένα και περισσότερος εξτρεμισμός. Ο κύριος Μίγιαν Μόν για δύο λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ζει μια πολύ μεγάλη κρίση το Ιράκ. Χθε εξελέγει ο προεδρο ε, της βουλη ε, Αυτό είναι μια καλή είδηση. Βέβαια, όπως πολλοί είπαν, δεν πρέπει να ξεχνάμε το σοβαρό κίνδυνο αποσύνθεσης ε, στη χώρα λόγω της ενοπλη επεμβαση του καλούμενου Ισλαμικού κρατου χθε όπως σα έλεγα, υπήρξε η συμφωνία για τον νέο πρόεδρο της Βουλής. Μια μικρή εξέλιξη θετική ε, που βλέπουμε μετά τις εκλογές ε, ε, της 30ης Απριλίου. Ελπίζω να έχουμε σύντομα το σχηματισμό μιας κυβέρνησης εθνικής ενότητας που να εκπροσωπεί ε, τα στρώματα όλα του πληθυσμού ή τέλο πάντων τα περισσότερα. Βλέπουμε πραγματικά μια διάσπαση του πληθυσμού που τίνει να καταστρέψει εντελώ οποιαδήποτε όνειρα του πληθυσμού για ειρήνη και ευημερία. Πρέπει να υπάρξει εθνική αλληλεγγύη, ε, ακαιρεότητα εδαφική, η τελο τα περισσοτερα βλεπουμε πραγματικα μια διασπαση του Ιράκ είναι κάτι αλληλεγγυη ακαιρεοτητα εδαφικη ανεξαρτησια του σημαντικό και στις 23 Ιουνίου το είπε και το Συμβούλιο Υπουργών ότι δεν θέλουμε σε καμία περίπτωση ε, τη διάσπαση της χώρας. Έχουμε λοιπόν αυτό αυτό το Ισλαμικό κράτος το οποίο και στο Ιράκ και στη Συρία σημειώνει μεγάλη ε, επιτυχία, προελάβνει ε, το ίσις δεν είναι μόνο τρομοκρατική ομάδα, είναι ένα στρατός, ε, τρομοκρατικός στρατός που θέτει σε κίνδυνο την παγκόσμια ασφάλεια. Θα πρέπει να συνεργαστούμε με όλες τις χώρες της περιοχής για να στηρίξουμε την εσωτερική σταθερότητα και την ενότητα της χώρας. Θα πρέπει επίσης η μεθόριος ε, Συρίας ε, και Ιράκ να μην γίνει Αφγανιστάν ε, της δεκαετίας του 90. Επίσης έχουμε εκατοντάδες χιλιάδες εκτοπισθέντες που βιώνουν τραγικές στιγμές. Και ολοκληρώνω κυρία Πρόεδρε τα τελευταία χρόνια επίσης έχει μειωθεί ο αριθμός των χριστιανών. Ε, όλα αυτά πρέπει να τα έχουμε υπόψη μας. Πρόεδρος, δέχεστε από τον κύριο Ορτασούνα ερώτηση, παρακαλώ. Μάλιστα. κύριο Ορτασούν. Ναι, πολύ ε, γρήγορα δύο ερωτήματα. Πρώτο ερώτημα, ποιο βαθμό ευθύνη αποδίδεται στον Χωσέ Μαρία Αφνάρ για τη σημερινή κατάσταση στο Ιράκ και δεύτερον, το Λαϊκό Κόμμα εξακολουθεί να πιστεύει ότι ήταν επιτυχία η επέμβαση στο Ιράκ. Απάντηση. Υπάρχουν πολλές αιτίε, κάποιες πιο μακρινές, κάποιες πιο ε, κοντινές για αυτή την κατάσταση στο Ιράκ. Ε, η επέμβαση στο Ιράκ έχει αποδειχθεί σε κάποια ε, στοιχεία τα οποία δυστυχώς εκ των αποδείχθηκαν εσφαλμένα. Ο κύριος Παπαδάκης τώρα έχει το λόγο για ένα λεπτό. Κύριε Πρόεδρε, η κατάσταση στο Ιράκ δεν είναι απλώς επικίνδυνη, αλλά είναι τραγικά επικίνδυνη. Και δεν αφορά μόνο το Ιράκ, αφορά τη Συρία, αφορά την Αίγυπτο, αφορά τη Λιβύη αποδεικνύεται ότι οι πολιτικές που ακολουθήθηκαν ήταν πέρα για πέρα λαθασμένες. δεν είναι τυχαίο ότι μόνο η τινησία οδηγήθηκε στην ομαλότητα στην περιοχή και υπάρχει αυτή τη στιγμή ένα καθεστώς αποσταθεροποίησης και δυστυχώς βλέπουμε ότι η αραβική άνοιξη έχει μετατραπεί σε ένα βαθύ αραβικό χειμώνα. είχαμε πολύ περισσότερες απώλειες ζωές το τελευταίο διάστημα και πολύ χειρότερες μορφές καταπίεσης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και καταπάτηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η απάντηση πρέπει να είναι ολοκληρωμένη από πλευρά τη Ευρώπη. Πρέπει να υπάρχει κοινή ευρωπαϊκή εξωτερική πολιτική η οποία να στηρίζεται σε πραγματικά δεδομένα και όχι σε ευσεβοποθισμού. Πρόεδρε, συνάδελφοι. Η ίσης έχει ανακοινώσει τη δημιουργία του χαλιφάτου. Ωρα, ο ριζοπαστικός Ισλαμισμός αποτελεί ένα από τις βασικότερες απειλές της, ε, του σύγχρονου πολιτισμού. Ο πόλεμος θα είναι πόλεμος των αξιών. Τα Δυτικά Βαλκάνια απειλούνται γιατί υπάρχουν μεγάλες μουσουλμανικές κοινότητες Ζούμε σε ειρηνική συμβίωση με τους ε, βουλγάρους μουσουλμάνους αδελφούς μας και δεν θέλουμε τέτοιες συγκρούσεις. Και η σημαία του χαλιφάτου ε, φάνηκε σε κάποιες συγκρούσεις στα Σκόπια την προηγούμενη εβδομάδα. Δεν θέλουμε να υπάρξει συνέχεια. Το ίσις ε, αναζητά νέους μαχητές σε μέρη όπως το Κάρντιφ και το νέο κύμα προσφύγων θα επιβαρύνει ιδιαίτερως την βουλγαρική οικονομία. Υπάρχει ψήφισμα του ECR και θα πρέπει να το εγκρίνουμε, να λάβουμε μέτρα για να ανταπεξέλθουμε στο κείμενο προσφύγων. Ευχαριστώ κύριε Αντακτούσον. Ευχαριστώ πρόεδρε. Καταρχάς θα ήθελα να πω ότι το σχέδιο νομοθετήματος ε, το υποστηρίζω. Ένα από τα μέρη που αναφέρονται είναι η πόλη Καρακός, η ασερική πόλη Καρακός, όπου χτίστηκαν εκκλησίες χριστιανικές ε, μισή χιλιετία πριν από τη, στη χώρα μου, την Σουηδία. Και αυτή τη φορά όταν ηχούν οι καμπάνες, δεν ηχούν για θρησκευτικούς σκοπούς, αλλά για να ειδοποιήσουν κατεπηγόντως τους πολίτες. Και λίγες μέρες μετά η πόλη είχε κενωθεί από χριστιανούς. Οι οικογένειες, οι συγγενείς των ατόμων αυτών που ζούσαν εδώ και γενιές ολόκληρες στην πόλη αυτή αναγκάστηκαν να τα παρατήσουν όλα και να φύγουν γιατί δεν μπορούσαν να μείνουν λόγω του μετόπου του ίσης στην Μοσούλη οι χριστιανικέ καμπάνες δεν αντίχησαν καθόλου την προηγούμενη Κυριακή. Για πρώτη φορά σε 600, 6.000 χρόνια δεν ε, έγινε, σε 1.600 χρόνια δεν ε, έγιναν θρησκευτικέ ε, λειτουργίε, χριστιανικές λειτουργίε. Και οι τζιχαστές, η τζιχάτ προτιμάει, προχωράει. Δεν μπορεί λοιπόν να παραμείνουμε απαθείς θα πρέπει να μπει ένα τέρμα στο Και θα πρέπει να προωθήσουμε μια κυβέρνηση εθνικής ενότητας. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επισκέφθηκε μια αερακινή κοινότητα την προηγούμενη εβδομάδα και υπογραμμίστηκε το θέμα αυτό της έλλειψης δημοκρατίας. Τα κράτη-μέλη θα πρέπει να υποστηρίξουν τις κοινότητες αυτές. Θα πρέπει πέρα από τα όρια των κομμάτων, των πολιτικών κομμάτων, να υποστηρίξουμε την αρρωγή αυτή μέσω του ψηφίσματος, αλλά θα πρέπει να τεθεί αυτό το θέμα και στην ε, ε ημερήσια διαταξή. Σας ευχαριστώ. Η ανομία, η διεφθαρμένη κυβέρνηση, η ασέβεια προς τα δικαιώματα των μειονοτήτων οδήγησαν στην κατάσταση αυτή που επικριτεί στο Ιράκ. Αυτό τα αναφέρει και το New York Times όπου ε, η κυβέρνηση Αλμαλίκη κάνει αυθαίρετες συλλήψεις σε Σουνίτες ε, Άραβες ε, και οι συνοπτικές εκτελέσεις έχουν γίνει το σύνηθες. Για χρόνια η διεθνής κοινότητα έχει πιέσει την κυβέρνηση των Σιτών να συμπεριλαμβάνει περισσότερο κόσμο από περισσότερε μειονότητε, αλλά χωρί αποτελέσματα. Υπάρχει ωστόσο μια ισχυρή ελπίδα με την ανακοίνωση ότι ένα Σουνίτη ορίστηκε πρόεδρο του Ιρακινού Κοινοβουλίου. Αυτό μάλλον δεν θα ωφελήσει και πολύ του αγωνιστέ Σουνίτε που έχουν διακηρύξει ένα, δημιουργία ενό Ισλαμικού κράτου εντό του κράτου. Και τώρα βλέπουμε ότι μπορεί να ξανασχεδιαστεί ο χάρτη τη Μέση Ανατολή με ε, απρόβλεπτες συνέπειες. Σε παρακαλώ να ολοκληρώσετε. Βέβαια, ε, δεν είμαστε αμέτωχοι σε όλη αυτή την κατάσταση και όπως και με τη σύγκρουση μεταξύ Ισραήλ και Παλαιστίνης θα πρέπει να γίνουν συγκεκριμένες και επίγουσες δράσεις από πλευράς Ένωσης. Ένα λεπτό έχει τώρα το λόγο η κυρία Φώτιγκα. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Το, το Ιράκ βρίσκεται στο χείλο του εμφυλίου πολέμου. Το ISIS έχει φτάσει πια στα προάστια της Ζαγδάτης. Ανίκανη κυβέρνηση που διχάζει το Ιρακινό κράτος είναι αυτή που φταίει για όλη αυτή την κατάσταση. καθώς και για την κατάσταση των χριστιανών εκεί που χρειάζονται την συντονισμένη προσπάθεια από πλευράς μας ώστε να υπάρξει μια κυβέρνηση ε, εθνικής συμφιλίωσης. Σας ευχαριστώ. Για δύο λεπτά η κυρία Γκαμπριέλα. Ε, καλά το είπατε το όνομά μου και στα βουλγάρικα, κυρία Πρόεδρε. Ε, η κατάσταση στο Ιράκ ε, και δεν είναι αυτό, είναι ιδιαίτερα ανησυχητικό. η, κατοχή από πλευρά ενό τμήματο του Ιράκ από μια τρομοκρατική ομάδα. Πρέπει να υπογραμμίσουμε ωστόσο την ευθύνη μια ε, πολιτική λύση ε, από πλευρά των ε, πολιτικών ευθυνών, ειδικά εκείνων που εξελέγησαν τον Απρίλιο στην Εθνοσυνέλευση. Θα πρέπει να αναλάβουν τι ευθύνε του απέναντι στο μέλλον και στου πολίτε. Είναι σαφέ ότι το Ιράκ δεν θα σηκώσει κεφάλι χωρί πραγματικό πολιτικό διάλογο και διαθρησκευτικό διάλογο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, δεύτερη μου παρατήρηση, είναι ότι θα πρέπει να συνεχίσει να δεσμεύεται και να βοηθά στα εκατομμύρια εκτοπισμένων ανθρώπων και στο 1,5 εκατομμύριο ανθρώπων που χρειάζονται ανθρωπιστική βοήθεια. Σήμερα και αυτό θα γίνει σε καλό, πρέπει να γίνει μάλλον σε καλό συντονισμό με τον ΟΗΕ, αλλά κυρίω προωθώντα τον πολιτικό διάλογο στην περιοχή. Τέλο, τελευταία μου παρατήρηση αφορά ε, κάτι που στο οποίο θα επιμείνω περισσότερο, ότι δηλαδή δεν μπορούμε να περιοριζόμαστε στο να αντιδρούμε μόνο στην ανθρωπιστική κατάσταση. Ήδη η περιφερειακή δυναμική στην περιοχή του Ιράκ θα πρέπει να έχει όλη μας την προσοχή. Η επεκτατική ατζέντα του τρομοκρατικής ε, ομάδας του ίσης δεν είναι απειλή μόνο για το Ιράκ τη Συρία, αλλά και ολόκληρη την περιοχή μέχρι και την Ιορδανία. Θα πρέπει επίσης να έχουμε υπόψη μας ότι οι ε, περιφερειακές συγκρούσεις μας απειλούν όπως και η σύγκριση ανάμεσα στους Ιήτες, στους Σουνίτες και τους Κούρδους. Θα πρέπει λοιπόν διαρκώς να παρακολουθούμε την κατάσταση σε αυτή την περιοχή που βρίσκεται στην πόρτα της Ευρώπης. Θα πρέπει ε, να γίνει ίσως και μια διάσκεψη ψηλού επίπεδου για να μην βρεθούμε σε μια κατάσταση όπου θα είμαστε δεμένα, δεμένοι, πιστάγκονα. Ευχαριστώ. Τώρα η κυρία Πύρη για ένα λεπτό. Ε, ευχαριστώ. Είναι πολύ ανησυχητικέ οι εξέλιξει στο Ιράκ και πραγματικά θα πρέπει να υπάρξει διεθνή αντίδραση. Η συνεχιζόμενη βία ε, έχει διώξει 1,2 εκατομμύρια ανθρώπους. Η ανθρωπαστική κρίση αυτή είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να γνωρίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι εικόνε που βλέπουμε μαζικών εκτελέσεων από τα τζιχαντιστικά Ακίνηματα είναι φρικτές και η κατάσταση είναι πάρα πολύ επικίνδυνη για όλη την περιοχή. Είναι πάρα πολύ σημαντικό λοιπόν η Ιρακινή κυβέρνηση μαζί με τις ε, ομάδες του πληθυσμού να προχωρήσει με την ε, ατζέντα της Εθνικής Συμφιλίωσης. Έγινε ένα πρώτο ενθαρρυντικό βήμα μέσω της εκλογής των Σουντιών στο Κοινοβούλιο. Θα πρέπει να, να παρακολουθήσουμε λοιπόν την κατάσταση από πλευρά της Ευρώπης γιατί ε, η έλξη των Ευρωπαίων ε, τσιχατιστών φαίνεται να αυξάνεται. Χρειάζεται συνεργασία για να καταπολεμήσουμε την ριζοπαστικοποίηση και την επιστροφή των ε, τσιχατιστών. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Τέλος η κυρία Μανέσκου για δύο λεπτά. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Τελευταία είμαστε μάρτυρες μια ε, σημαντική επιδείνωση της κατάσταση στο Ιράκ με βίαιες επιθέσεις ε, κατά πολιτών που είναι θύματα της τρομοκρατίας. Είναι λυπηρό το γεγονό ότι η Ιρακινή κυβέρνηση ε, απεδείχθη ανίκανη να προφυλάξει και να υπερασπιστεί τους πολίτες από τους τρομοκράτες. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλοι σύμμαχοι πρέπει να ε, επηρεάσουμε, αλλά αυτό μπορούμε να το πράξουμε μόνο εάν ε, και οι ηγέτες ε, της χώρας ασχοληθούν με το πρόβλημα σοβαρά και αποφασίσουν να βάλουν πρώτη προτεραιότητα τη σταθεροποίηση της χώρας. Ήταν καταστροφική η πολιτική του Αλμαλίκη που έφερε σε ανταγωνισμό τις διάφορες εθνοτικές και θρησκευτικέ ομάδες. Εμείς θέλουμε να στηρίξουμε και στο μέλλον το Ιράκ με ανθρωπιστική βοήθεια. Είναι σημαντικό να δείξουμε την αλληλεγγύη μας, να δετρανώσουμε την αλληλεγγύη μας με τον Ιρακινό λαό. Και να μην ξεχάσουμε ότι όπως έχει αποδείξει η ιστορία ο στρατιωτικός ε, επεμβατισμός μόνο προβλήματα δημιουργεί. Αυτό που βλέπουμε είναι ιστορικές στιγμές για την ε, χώρα του Ιράκ αλλά και για την ευρύτερη περιοχή. Θα πρέπει οι ηγέτες ε, της χώρας να ε, υπερκεράσουν τις θρησκευτικέ διαφορές και να οραματιστούν ένα κοινό μέλλον για το Ιράκ. Η διεθνής κοινότητα μπορεί επίσης να φέρει την ε, ειρήνη και τη σταθερότητα. Και θα πρέπει στην κυβέρνηση να είναι τόσο συνήθως όσο και σύντες. Με το διάλογο ε, μπορεί να δημιουργηθεί ένα ισχυρό Ιρακινό κράτος. Το Ιράκ αυτό που χρειάζεται σήμερα είναι μια νέα κυβέρνηση. Μια κυβέρνηση της οποίας θα ηγείται ένας διαφορετικό πρωθυπουργό, ένα άλλο πρωθυπουργό, όχι ο Αλμαλίκη, ένα πρωθυπουργό που θα εκπροσωπεί όλου του Ιρακινού πολίτε, ανεξαρτήτω ε, εθνοτική ή θρησκευτική προέλευση. Περνάμε στη δικασία Catch the Eye, προσέλκυση προσοχή του πέντε τη. Ο κύριο Τηλιανίδη είναι ο πρώτο. Ε, Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Επιτρέψτε μου να θέσω κάτι διαφορετικό αλλά πάρα πολύ σχετικό με τη συζήτησή μας. Η ανησυχητική κατάσταση στο Ιράκ και στη Μέση Ανατολή θα σήμαινε τεράστιες γεωπολιτικές αλλαγές συμπεριλαμβανομένης και της αλλαγής ενδεχομένως των συνόρων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και η διεθνής κοινότητα δεν ήταν δυνατόν να παρέμβουν στην ευρύτερη περιοχή με επικοδομητικό τρόπο. Όλα αυτά τα περιστατικά θα υπονόμευαν περαιτέρω την ασφάλεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ιδιαίτερα στην ενεργειακή ασφάλεια. Είναι λοιπόν ε, καιρός να ξανασκεφτούμε την ενεργειακό εφοδιασμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι καιρός να αναζητήσουμε ε, διαδρομές ε, και εταίρους πιο ασφαλείς για τον ενεργειακό εφοδιασμό. Αν θέλετε να ολοκληρώσετε, λέει η Πρόεδρος, θα πρέπει να κοιτάξουμε πώς μπορούμε να εκμεταλλευτούμε τα αποθέματα στην ε, Μεσόγειο. Αυτό θα είναι πραγματικά κάτι σημαντικό και θα πρέπει να το θέσουμε ο κύριος Φεραίρα. για ένα λεπτό, λέει η Πρόεδρος. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πριν από κάποια χρόνια ο στρατηγός ε, Πίτερς ε, δημοσίευσε έναν χάρτη παράξενο που μας παραξένευσε. Ήταν ο νέος χάρτης για τη Μέση Ανατολή. Μετά προοπτική των χρόνο που πέρασαν και τα ε, τελευταία συμβάντα αποκτούν όλα νόημα με βάση το χάρτη του στρατηγού Πίτερς. Είναι μια παλιά τεχνική περιελιστικής κατάκτησης της ε, και Βασίλευε ε, η χρήση των ε, των ε, πληρωμένων στρατιωτικών, των μισθοφόρων, ε, καθώς και η χρήση των ε, μισθοφόρων και στη Συρία που έσπηραν το χάος. Αυτές οι προσπάθειες σκοπεύουν σε όλες τις χώρες που τις τελευταίες δεκαετίες έχουν αποτελέσει τις κλίνες όλων των, μάλλον τα φυτόρια όλων των υπηρελιστικών προθέσεων στην περιοχή η περίπτωση της Συρίας αλλά και του Ιράκ αλλά και ολόκληρης Μέσης Ανατολής δεν είναι τυχαία. Ευχαριστώ για ένα λεπτό κύριο Νικολάσιτς. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Θα ήθελα και εγώ να πάρω το λόγο για την κατάσταση η οποία είναι ιδιαίτερο ανησυχητική και προκαλεί παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο βόρειο τμήμα του Ιράκ δημιουργήθηκε ένα χαλιφάτο όπου ισχύει ο νόμος της Αρίας και αυτό τι σημαίνει θάνατος στους αλόπιστους. Αυτά λοιπόν είναι τα γεγονότα. Σε πρώτο βήμα ξεκίνησαν ε, να καταπολεμούν τους ε, αδερφούς τους. Δύο ομάδες λοιπόν, οι Σουνίτες, οι Σίτες και ε, οι μεν πολεμούν τους Αυτό που είναι ιδιαίτερα ανησυχητικό είναι ότι η κατάσταση αυτή μας οδηγεί σε επιδείνωση της κατάστασης των χριστιανών, οι οποίοι ζουν εκεί εδώ και χιλιάδες, ε, πάνω από χίλια χρόνια. Και αυτό λοιπόν είναι καθήκον μας, είναι καθήκον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να προσπαθήσει τα δικαιώματά τους. Είναι σκανδαλώδες και κλείνω το ότι το Συμβούλιο βρίσκεται εδώ, αλλά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν παρευρίσκεται. Για ένα λεπτό, ο κύριος Εφρίτς, λέει η Πρόεδρος. Thank Σας ευχαριστώ. Θα ήθελα να επιδείξουμε μεγάλη προσοχή, γιατί το πρώτο ένστικτό μας θα ήταν να παρεμβούμε. Και με καλούς σκοπούς συχνά, αλλά για πολλές δεκαετίες η κατάσταση στη Μέση Ανατολή επιδεινώνεται όλο και πιο πολύ από την παρέμβαση του δυτικού κόσμου. Και η δική μου χώρα ε, ε, έδρασε με τα αποψεύματα του Τόνι Μπλερ. Έχει αίμα στα χέρια του. Και γι' αυτό λοιπόν βρισκόμαστε στην τρέχουσα κατάσταση. Ας διδαχθούμε λοιπόν από τα παθήματα του παρελθόντος. Δεν είναι δυνατόν να είμαστε εμείς η αστυνομία του, όλου, του κόσμου. Να βοηθήσουμε, δεν λέω, που μπορούμε, αλλά σας παρακαλώ για την ειρήνη, ας μην προσπαθούμε πάντα να παρεμβαίνουμε Ας μην προσπαθούμε πάντα να μπλεκόμαστε, γιατί σε κάποιες περιπτώσεις είναι καλύτερα να σεβόμαστε την εθνική ανεξαρτησία και να αφήσουμε τον κόσμο να ζει σύμφωνα με τις δικές του επιλογές. Και τώρα το λόγο έχει ο κ. Κίρτσος για ένα λεπτό. Ε, νομίζω ότι το Ιράκ έχει μπει στην τελική φάση της διάλυσης και είναι μια τεράστια απόσταση που έχει καλυφθεί με την αρνητική έννοια του όρου, διότι να θυμίσουμε ότι υπήρχε μια φιλοδοξία για το λεγόμενο nation building μια σύγχρονη δημοκρατία θα δημιουργούνται εκεί και τώρα έχουμε ένα αιματηρό χάο. πιστεύω ότι αν είχαμε περισσότερη ευρώπη θα είχαμε λιγότερα λάθη και στην περίπτωση του ιράκ. εάν, δεν διστάζαμε να αποκτήσουμε κοινή εξωτερική πολιτική εάν δεν διστάζαμε να αποκτήσουμε κοινή αμυντική πολιτική θα είχαμε παρεμβάσει προ τη σωστή κατεύθυνση. Μα φοβίζει το κόστο, αλλά τελικά δεν μπορούμε να το αποφύγουμε διότι η κατάρρευση του ιράκ μπορεί να οδηγήσει σε ενεργειακή κρίση που θα έχει τεράστιο κόστος μπορεί να οδηγήσει στην ενίσχυση του ιράν και στην κλιμάκωση της αντιπαράθεσης με το ισραήλ που και αυτό θα έχει συνέπειες μπορεί να οδηγήσει σε ένα νέο κύμα προσφύγων που θα είναι εξαιρετικά δαπανηρό μπορεί να οδηγήσει ακόμα και στην ενίσχυση των φανατικών ισλαμιστών και την αποσταθεροποίηση των ε, κυβερνήσεων στον αραβικό κόσμο. επομένως ό,τι και να κάνουμε έχουμε ένα λογαριασμό μπροστά μα η περισσότερη ευρώπη είναι η οικονομικότερη προοπτική. Είχα και τον κύριο Γλέζο στον κατάλογό μου. Τον ξέχασα. Άρα έκτο ο και τελευταίο. Ο κύριο Γλέζο, ένα λεπτό. Πριν από 71 χρόνια, αγαπητοί συνάδελφοι, συνήλθαν στη Γιάλτα οι λεγόμενοι τρει μεγάλοι. Ο Ρούσβελτ, ο Τσόρτσιλ και ο Στάλιν και ανακοίνωσαν εκφράζοντας τις επιθυμίες των λαών ότι μετά τη λήξη του πολέμου θα καταργηθεί η απεικιοκρατία, θα υπάρξει αυτοδιάθεση των λαών, σεβασμός των μειονοτήτων και ατομικά δικαιώματα. Ας μην στρωθο... στρουθοκαμιλίζουμε. Σήμερα θέλουμε δεν το θέλουμε αυτά τα εξαγγελθέντα από τους τρεις δεν υπάρχουν στην πραγματικότητα. Υπάρχει πρόβλημα αυτοδιάθεσης λαών, υπάρχει πρόβλημα αυτοδιάθεσης των Κούρδων και πώς να το κουβεδιάσουμε όταν υπάρχει η Ιρλανδία που δεν έχει αποκτήσει ολόκληρη την ανεξαρτησία της, υπάρχουν οι Βάσκοι, υπάρχουν οι Καταλανοί, υπάρχουν οι Βορειοπυρώτες επιτέλους θα αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα ναι ή όχι. Σας ευχαριστώ. Ολοκληρώνεται με τον κύριο Κλέζο η διαδικασία Catch the Eye και θα δώσω τώρα τον λόγο στον κύριο Ντελαβέντοβα. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ όλους τους ευρωβουλευτές που πήραν τον λόγο στη διάρκεια αυτή τη ειλικρινούς και εις βάθος που μόλις ολοκληρώθηκε. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει την πρόθεση και νομίζω πως και εσείς δικαίως το ζητήσατε να συζητήσει το θέμα λοιπόν του Ιράκ. Συζητήθηκε στο Συμβούλιο της 24ης Ιουνίου. Μια νέα συζήτηση προβλέπεται για το θέμα του Ιράκ την επόμενη εβδομάδα στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων ε, που έχει προβλεφθεί για τις 22 Ιουλίου. Ανάμεσα στα θέματα τα οποία εσείς αναφέρατε ε, είναι η κοινή δέσμευση δηλαδή της ενότητας και της ακεραιότητας ε, της εδαφικής του Ιράκ. Αυτό τα αναφέρεται ως βασικά στοιχεία για να οικοδομηθεί μια ευημερία που να είναι προς όφελος όλων των πολιτών και που θα προωθεί τη σταθερότητα στην περιοχή. Δεν διαφεύγει κανενός βεβαίως η σοβαρότητα και η δραματικότητα της κατάστασης Οι αρχικές ε, παρεμβάσεις του κυρίου ε, Νότ και, του κυρίου, και της κυρίας Γκόμες ε, ανέφεραν στήριξη σταθερή και προώθηση μιας κρατικής και ενωτικής διακυβέρνησης μέσα στο πλαίσιο του συντάγματος ή εν πάση περιπτώσει μια διακυβέρνηση που να επιτρέπει να συνεχιστεί η διαδικασία μετάβασης προς την δημοκρατία. Ε, το θέμα αυτό βέβαια είναι ένα θέμα που ιστορικά αλλά και αυτή τη φορά ε, προκαλεί τα αισθήματα ολόκληρη της Ευρώπης ε, και αφορά την ελευθερία των χριστιανών πιστών που βρίσκονται στην περιοχή. Και γι' αυτό το λόγο ε, θα χρησιμεύσει μια νέα Ιρακινή κυβέρνηση η οποία θα είναι νόμιμη και θα συμπεριλαμβάνει όλες τις συνιστώσεις και για αυτό το επίπεδο, σε αυτό το επίπεδο κινούμεθα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ήθελα μάλιστα να μιλήσω για δύο, συγκεκριμένες, ε, δύο συγκεκριμένα αιτήματα που γίνονται σε σχέση με το θέμα των χημικών όπλων η Πηγές ε, της κατασκοπίας επιβεβαιώνουν ότι δεν πρόκειται για ε, όπλα τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Βέβαια, μέσα σε αυτό το χάος είναι απαραίτητο να παραμένουμε στα γνωστά στοιχεία και στα επιβεβαιωμένα στοιχεία. Τώρα όσον αφορά τις ε, κατηγορίες προς την Τουρκία όσον αφορά τη χρηματοδότηση του ΙΖΙΛ ε, θα πρέπει να διατηρούμε μια διαφορά και να κάνουμε μια σαφή διάκριση ανάμεσα στις υποψίες, τις φήμες και στα ε, γεγονότα, τα στοιχειοθετημένα και ε, τις χρηματοδοτήσεις που ίσως να προέρχονται από ακραίους ιδιωτικούς φορείς και, την κυβέρ... και χωριστά την κυβέρνηση της Τουρκίας. Πρέπει η διάκριση δηλαδή να γίνεται ανάμεσα στην κυβέρνηση της Τουρκίας και τις ιδιωτικές ε, χρηματοδοτήσεις. Πάντως θα πρέπει να αποφύγουμε τη χρηματοδότηση του Ίζιλ και άλλων τρομοκρατικών ομάδων. Τέλος θα ήθελα να εκφράσω την εκτίμησή μου που νομίζω θα συμφωνήσετε κι εσείς για την εξαίρετη δουλειά της αντιπροσωπείας μας στην Βαγδάτη. Οι συναδελφοί μας στο Ιράκ εξακολουθούν να προσφέρουν πολύτιμη υπηρεσία σε συνθήκες εξαιρετικά δύσκολες. Ευχαριστώ. Σα ευχαριστώ. Λάβαμε έξι προτάσει ψηφίσματο για να ολοκληρωθεί αυτή η συζήτηση που κλείνει τώρα και η ψηφορία θα γίνει αύριο στι 11. Σα ευχαριστώ. Σύμφωνα με την ημερήσια διάταξη, θα ακούσουμε τώρα τη δήλωση τη Αντιπροέδρου τη Επιτροπή Υπέρ τη τη Ένωση για θέματα εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλεια σε σχέση με την κλιμάκωση τη βία μεταξύ Ισραήλ και Παλαιστίνη. Και ξαναδίνω το λόγο στον κύριο